colleagues, uh, I was suggested that we should start the meeting and uh, our να ξεκινήσουμε και όπου να θα φτάσει και ο πρόεδρος. Ελπίζω σύντομα να είναι εδώ μαζί μας πάλι. Λοιπόν, Καλημέρα σε όλους σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την έγκριση της μερισίας διατάξεως. Να σας πω ότι τα σημεία 9 και 10, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας σχετικά με την απλούστευση στην έκδοση θεωρήσεων και Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοκρατίας, Αρμεν... Αρμενίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια ε, αναβάλλονται μετά από αίτημα της εισηγητρίας Επομένως ε, θα εγκρίνουμε την τροποποιημένη ημερήσια διάταξη. Πολύ ωραία. Στις ανακοινώσεις του Πρόεδρου δεν έχουμε τίποτα. Πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης ε, της 9ης και της 10ης Οκτωβρίου του 12 και εδώ δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια και παρατηρήσεις και επομένως να μελετήσουμε το επόμενο ζήτημα, δηλαδή ε, νομοθετικές διαδικασίες Ε, σχετικά με τον έκτο τριμερή διάλογο για τους εποχικούς εργαζόμενους. Ο κύριος Μωράες, ο εισηγητής, μπορεί να μας πει δύο λόγια όσον αφορά ε, την ε, κατάσταση. Είχαμε λοιπόν τον πέμπτο διάλογο για τους εποχικούς, τριμερή διάλογο για τους εποχικούς εργαζόμενους και παρότι δεν επιτύχαμε συμφωνία πιστεύω ότι αυτός ο τριμερής διάλογος υπό Ιρλανδική Προεδρία ήταν πάρα πολύ θετικός ε, να ευχαριστήσουμε και όλα την Προεδρία, την Ιρλανδική Προεδρία, γιατί προχωρήσαμε πολύ πάνω σε συγκεκριμένα ε, ζητήματα κεντρικού ενδιαφέροντος. Το θέμα των εποχικών εργαζόμενων είναι ευαίσθητο γιατί είναι η μόνη ε, επίσημη μορφή, νόμιμη μάλλον μορφή μετανάστευσης για ε, εργάτες και εργαζόμενους ε, χωρίς γνώσεις. Ευαίσθητα λοιπόν θέματα, επί των οποίων έχει γίνει πρόοδος, δυστυχώς όμως δεν επιτεύχθη η συμφωνία. Ευελπιστώ πάντως ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση, να ολοκληρώσουμε δηλαδή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε τριμερή διάλογο την 8η Ιουλίου και ε, ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε ε, να έχουμε μια τελική λύση γιατί ξέρετε έχουν κουραστεί και όλοι οι εμπλεκόμενοι ε, στις 8 Ιουλίου ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Να ευχαριστήσω πάντως ιδιαιτέρως ήθελα την Ιρλανδική Προεδρία και τους και τους υπαλλήλους γιατί δούλεψαν πάρα πολύ. Παρότι δεν φτάσαμε, λέω, σε τελική συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μωράης. έκθεση HEG σχετικά με τις, προ... σχετικά με τις προμήθειες. Ε, η Κορεπέρα, από ό,τι μαθαίνω, χτες ενέκρινε το κείμενο ε, και τις... Ε, συγγνώμη για το θέμα των προδρόμων ουσιών. Η συγγήτρια δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά θα ήθελα να τη συγχαρώ, καθώς επίσης και όλους τους σκιώδεις για τα καλά αποτελέσματα. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 6 της ημερησίας διατάξεως, χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών, δεδομένα PNR δηλαδή, ο κύριος Κύρκοπ. Έχουμε μία πρόταση η οποία εκκρεμεί από το 2011. Επανειλημμένα συζητήθηκε το θέμα ε, στην ε, ε, Επιτροπή. Θέματα όπως ας πούμε η αναλογικότητα, η νομική προστασία, δικαιώματα πολιτών κτλ. μας απασχόλησαν εδώ. Ε, λοιπόν, έγινε μια τελική έκθεση η οποία έφτασε στην Ολομέλεια σύμφωνα με τον, ε, κανόνα, τον άρθρο 275 του ιστορικού κανονισμού ε, μετά από απόρριψη της Ολομέλειας ξαναήρθε το θέμα στην Επιτροπή και δίνω τον λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα των ταξιδιωτών στις αεροπορικές εταιρείε και τα δεδομένα τους. Είμαστε εδώ επειδή σε σχέση με το Κοινοβούλιο αποφάσισε να επανέλθουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα συμβιβασμό αντί να απορριφθεί αυτή η πρόταση. Αυτή φυσικά είναι και η πρόθεσή μου. Και από εδώ φυσικά ελπίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με επικοδομητικό τρόπο για αυτό το θέμα. Πρόεδρε, εσείς προηγούμενα σκιαγραφίσατε τα κυριότερα θέματα ως παιδεία. Ελπίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια συμφωνία. Όλοι θα έχετε συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα αυτού του φάκελου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θεμελιωδών δικαιωμάτων των ταξιδιωτών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ένα θέμα που έχει τεράστια εμβέλεια και που δημιούργησε ειδική επιτροπή το σώμα, την Επιτροπή Κρίμ για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού και θα ακούσουμε σε σχέση με διάφορους που θα μιλήσουν για την οδηγία, για την προστασία δεδομένων και που έγινε λόγος ε, και για ένα τέτοιο σύστημα και την αναγκαιότητά του Α, τέτοιου είδος ε, ανησυχίες και τοποθετήσεις τις κατανοώ. Γι' αυτό είναι όμως σημαντικό να έχουμε σαφές νομικό πλαίσιο από πλευράς της Ευρώπης και δεδομένα όσον αφορά τα δικαιώματα, ώστε οι επιβάτες ε, για τα δικαιώματά τους σε σχέση με αυτό το θέμα διαβίβασης δεδομένων που δεν ρυθμίζεται αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό επίπεδο και όπου είδαμε σαφώς ε, τυχαία συστήματα να αναφύονται σε τακτά διαστήματα, συγκυριακά, αυτή η οδηγία αντιμετωπίζει την χρήση των προσωπικών δεδομένων των ταξιδιωτών με τρόπο που δεν καλύπτεται από την οδηγία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, που πήρε αρκετό χρόνο για να υιοθετηθεί κατά το παρελθόν. Ελπίζω ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να μας επεξηγήσει την αξία των δεδομένων αυτών και γιατί είναι θεμελιώδου σημασία ένας μεγαλύτερος αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα να θέσουν σε τάξη τα συστήματα αυτά σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξει επικοδομητική προσέγγιση ώστε να προαχθεί αυτό το φατοφυλάκιο. Μα έδωσε σαφή εντολή η Επίτροπη για να δούμε αυτό το θέμα και να το εξετάσουμε με υπεύθυνο τρόπο. Προσέφερα στους συνεισηγητές και σκιώδεις εισηγητές μια ευκαιρία να μπορέσουμε να ε, βρούμε λύσεις και ελπίζω ότι θα επανέλθουμε σύντομα για να συζητήσουμε πώς ακριβώς ε, θα πορευτούμε στο μέλλον. Γι' αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα τη σπουδαιότητα αυτού του ζητήματος προς ε, το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων ταξιδιωτών και πολιτών. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Κίρκο. Άλλος που θα ήθελε να παρέμβει, παρακαλώ. Όχι, κανείς. Η κυρία Ρομέρο. Ναι, παρακαλώ κυρία Ρομέρο Λόπε, έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Με ικανοποίηση για την έκθεση της ε, παρουσίασης της θέσης ε, της ε, Επιτροπής. Είμαι εγώ σκιώδης εισηγήτριας από πλάστον των σοσιαλδημοκρατών η πρόταση λοιπόν του κύριου Κέρκοπ πλησιάστε το μικρόφωνο. Ναι, μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα υπό το πρίσμα ότι πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο να εκπονώντας επεξεργαζόμενη αυτή την πρόταση είναι μια περίπλοκη πρόταση και η κατάσταση επιπλέον μέσα στην οποία διεξάγεται αυτή η συζήτηση είναι περίπλοκη και ακαθόδη συζήτηση παρακολουθούμε αυτή τη συζήτηση με την οδηγία προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων που είναι σημαντική υπόθεση και για όλα αυτά πιστεύω ότι αυτή μπορεί να είναι μια ευκαιρία για μας ώστε να συνεχίσουμε τη συζήτηση σε αυτό το θέμα που δεν έχει αποσαφινιστεί απόλυτα ακόμα με κανένα τρόπο. Και τώρα για τους λόγους ε, για την απόρριψη σε σχέση, όχι γι' αυτό, αλλά επειδή υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν προσθεθεί επιπλέον και έχουν υπαρθεί σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο ε, εντάσσεται στην προστασία προσωπικών δεδομένων και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Υπάρχει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και δεν πρέπει να διαραγεί αυτό και είναι προφανέ ότι για να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί ένα τέτοιο κλίμα εμπιστοσύνη πρέπει να υπάρξει αποσαφήνιση και διευκρινήσει σε πολλά θέματα για τα θεμέλια επί των οποίων θα βασίσουμε τι προτάσει μα για την ασφάλεια και την καταπολέμηση του εγκλήματο. Γι' αυτό λοιπόν ενδιαφέρον θα ήταν πιστεύω να έχουμε και μια άλλη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση προσπαθώντας να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για αυτό το θέμα γιατί αυτή είναι η θέση της ομάδας μας και την γνωρίζει ο κύριος Κερκόπ σε σχέση και με τις τροπολογίες. Να συνεχίσουμε τη δουλειά, διότι πολλά σημεία πρέπει να αποσαφινιστούν που δεν έχουν αποσαφινιστεί και είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά προς αυτή την αποσαφήνιση. Ευχαριστώ. Frau Ernst, bitte. Κυρία Ernst, παρακαλώ. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το ότι η συζήτηση αυτή εγγράφηκε και ξεκινά έτσι και σε εμά σήμερα και δικό μας αίτημα είναι και υπήρξε ανταπόκριση όσον αφορά αυτό. Είχαμε ακριβώς στραφεί σε σχέση με τη συζήτηση να δούμε πόσο θα υπάρξει συνέχεια από αυτού του θέματος. Και με τα πιο πρόσφατα σκάνδαλα τα οποία αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε που από κυβερνήσεις τις ίδιες προκλήθηκαν και διεξήχθησαν και ε, είχαν αναπτυχθεί, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να δούμε πώς τα προσωπικά δεδομένα θα διασφαλίζονται όσον αφορά τους πολίτες της Ευρώπης. Πράγμα που είναι αναγκαίο για να διασφαλίζονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα και να υπάρχει ασφάλεια. Ασφάλεια να ανταποκριθούμε στα ε, αιτήματα για τη διασφάλιση ενός πλαισίου που θα ε, κατοχυρώνει την ασφάλειά μας. Πρέπει να διεξαχθεί λοιπόν μια συζήτηση, να γίνουν διαβήματα και βήματα, προτού όμως συνεχίσουμε τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα PNR, είναι κατεπηγόντως αναγκαίο να κάνουμε μια κοινή συνάντηση με όλους τους εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές για τα θέματα εκείνα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή τον κανονισμό προστασίας δεδομένων, την οδηγία προστασίας δεδομένων τα, την Ευρωπαϊκή Συμφωνία προς, ε, Ανταλλαγής ή Διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων και Ονομάτων Επιβατών, σε όλα αυτά πρέπει να συζητήσουμε καταρχήν ποια, ποια διασύνδεση υπάρχει μεταξύ αυτών των θεμάτων ποια επί της ουσίας ε, αλληλουχία υπάρχει και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα στη συνέχεια. Νυφάλια και ήρεμα πρέπει να τα, συζητήσουμε με επαρκές χρονικό όριο στη, ε, πλαίσιο στη διάθεσή μας. Πρέπει επίσης να αποσαφηνίσουμε τι αληθεύει και τι όχι, ποια είναι τα γεγονότα και δεδομένα τι συμβαίνει σε σχέση με τα κράτη-μέλη, κατά πόσον υλοποιούν πρώτον τέτοιου είδους ε, συμφωνίες ή αιτήματα για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων ταξιδιωτών και τι γίνεται σε σχέση με τα επιχειρήματα αυτών των κρατών μελών που ακολουθούν μια τέτοια τάση ή κατεύθυνση. Θα θέλαμε ακριβώς να γνωρίζουμε τι συμβαίνει ώστε να μπορούμε με βάση αυτά τα δεδομένα να συζητούμε εδώ και όχι να λέμε κατονομάζοντας κάποιες χώρες ότι η μία ή η άλλη χώρα κάνει κάτι. Αυτό δεν επαρκεί και επανειλημμένα σε σχέση με τις αρχές ε, προστασίας δεδομένων να έχουμε και την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Δεδομένων με την οποία θα έρθουμε σε επαφή και θα συζητήσουμε πρέπει να υπάρξει επαρκής χρόνος για αυτή την ε, ε, σημαντική απόφαση που πρέπει να λάβουμε. Αυτή είναι η πρότασή μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Για το ένα, καταρχήν θέλω να χαιρετήσω πρώτον ότι ο εισηγητής εδώ για άλλη μία φορά κάνει την προσπάθεια να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, να συνεχίσουμε τη συζήτηση για αυτό που κάπως, ας το πω έτσι, ε, δεν έχει ακολουθήσει την σωστότερη διαδικασία και λόγω της ουσίας και λόγω άλλων θεμάτων που δεν καταφέραμε πλειοψηφικά να έχουμε κάποια θεμέλια μέσα στα οποία θα τα εντάσαμε αυτά, ενιαίο πλαίσιο για παράδειγμα. Για αυτά που αναφέρθηκαν, Δεν ήθελα και εγώ σύντομα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία. Με βάση αυτά τα σκάνδαλα για την συλλογή προσωπικών δεδομένων από κάποιες υπηρεσίες μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια είναι η μεγάλη αξία μιας, ενός ρυθμιστικού πλαισίου. Αυτό το σκάνδαλο για τα προσωπικά δεδομένα στην Αμερική συνέβη επειδή δεν υπάρχει ρύθμιση για αυτά τα, θέματα και είναι κατεπήγον τώρα πιστεύω να υπάρξει μια ρύθμιση, ε, ένα κανονιστικό πλαίσιο. Για τα θέματα τα οποία προαναφέρθηκαν δεν μπορώ εγώ να δω κατά πόσον αυτό, αυτά είναι τα πιο ε, εύθετα. Τώρα, σε ποια πεδία, σε ποια πλαίσια θα κινηθούμε δεν έχει καμιά σχέση με την ίδια την οδηγία ή την ίδια την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αυτά τα θέματα εκεί δεν μπορούν να επιληθούν σε σχέση με τα δεδομένα PNR για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά πρέπει να επιληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια και να υπάρξει λέξη ειδικό νομοθέτημα. Σε αυτή την οδηγία, σε αυτόν τον κανονισμό δεν κανονίζουμε κατά ποια περίοδο θα μπορούν να αποθηκευθούν τέτοιου είδους δεδομένα, ούτε ρυθμίζονται ποιες πτήσεις καλύπτονται. Κάποιες αρχές μόνο καλύπτονται και αναφέρονται. Και αυτές πρέπει να μεταφερθούν στην οδηγία για τα PNR της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό αυτή η αλληλοδιασύνδεση, η αλληλουχία δεν είναι κάτι το πολύ σημαντικό για μένα. Δεν είναι δεδομένο. Μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, αλλά επί της ουσίας δεν θα άλλαζε και τόσα πολλά πράγματα. Το χαιρετίζω κατά τούτο λοιπόν αν μπορέσουμε στην περαιτέρω συζήτηση ίσως να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς που θα τύχουν πλειοψηφικά έγκρισης, διότι οι εξελίξεις στα κράτη-μέλη σε αυτά τα θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και PNR συνεχίζεται η συζήτηση αυτή, επειδή επιτρέπεται, επειδή δεν υπάρχει ένα αριθμιστικό πλαίσιο και στη συνέχεια θα είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά να τα μπορέσουμε να τα εντάξουμε σε ένα ενίο πλαίσιο. Γι' αυτό πρέπει το δυνατό πιο γοργά να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Ιντφέλτ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σύντομα κι εγώ γιατί θα ήθελα στα διαδικαστικά να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πολλή δουλειά έγινε ήδη επί της ουσίας και είμαι βέβαια ότι πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν και να βελτιωθούν για το ζήτημα της ουσίας. Από την πρώτη μέρα ευθύ εξ αρχής δύο παρατηρήσεις έκανα και παραμένω και εμένω σε αυτές τις παρατηρήσεις. Πρώτον, αν πούμε ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή οδηγία για να εναρμονίσουμε το πλαίσιο των εθνικών δεδομένων σήμερα, τότε θέλω να μου δοθούν πληροφορίες για αυτά τα εθνικά πλαίσια σήμερα. Σήμερα και τα ζητήσαμε αυτά, εδώ και χρόνια τα ζητάμε, δεν τα ζητάμε σήμερα μόνο ότι 16 ε, χώρες που έχουν τέτοια προγράμματα, πολύ ωραία λοιπόν, να μας δοθούν λεπτομέρειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Δεν είναι υπερβολικό ως αίτημα αυτό πιστεύω. Δεύτερον, γνωρίζω ότι κάποιοι διαφωνούν, αλλά πιστεύω και από την πρώτη μέρα το έλεγα ότι διασυνδέεται αυτό με την οδηγία προστασία προσωπικών δεδομένων. Δεν έχει κανένα νόημα θα έλεγα να δημιουργήσουμε ένα πεδίο για τη συνεργασία δικαστικών αρχών και αστυνομικών αρχών. Είμαι υπέρ εγώ να υπάρξει τέτοια συνεργασία και να βελτιωθεί αλλά να βασίζεται σε μια ρύθμιση για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων. Δεν πρέπει την προστασία προσωπικών δεδομένων για κάθε διάταξη οδηγία ή κανονισμό να την επαναδιαπραγματευόμαστε κάθε φορά εκ νέου. Να έχουμε για παράδειγμα για τους ταξι, τα ταξιδιωτικά στοιχεία των επιβατών προς τη ΣΥΠΑ, μία ρύθμιση για άλλα θέματα, άλλες ξεχωριστές ρυθμίσεις. Δεν είναι σοβαρός τρόπος ε, να ρυθμίζουμε τα πράγματα αυτό. Ξέρω ότι είπαν πολλοί, εντάξει να διασυνδεθούν τα δύο. Θα πάρει χρόνια όμως αυτό. Πολλά αποκαλύπτει. Ε, θα το δεχτούμε αυτό. Ήδη βλέπουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει πρόθεση να υιοθετήσει λοιπόν την οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό ανατρέπει και αλλάζει όλη τη στρατηγική και όλα τα δεδομένα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως σύνολο. Εμεί με αυτή την υπόθεση εργαζόμαστε, ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του το Συμβούλιο και θα μπορέσει αυτό να προωθεί μέχρι ότου δηλωθεί ότι δεν ισχύει αυτό. Ε, τουλάχιστον να μα το πει δημόσια λοιπόν το Συμβούλιο. Μέχρι νεοτέρας λοιπόν, εγώ θα υποθέτω ότι θα εγκριθεί, πρόκειται να εγκριθεί η Οδηγία προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Και έχω πρόθεση να εργαστώ κι εγώ για την οδηγία για τα, τα PNR στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω και εγώ από πλευράς μου ότι είμαι κάπως απογοητευμένος ακόμα για το ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ψήφιζε με σαφήνεια για την επαναπομπή στην ε, Επιτροπή ή την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής και μετά στη συνέχεια αποσύρθηκε από την ολομέλεια αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας, νομίζω, στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πρέπει να εμείνουμε και να επιμείνουμε στις αποφάσεις μας. Τώρα, για το θέμα ουσίας. Ξέρετε ότι έχω προαναγγείλει πολλές φορές ότι υπάρχουν σημαντικότατες ε, συνταγματικές επιπτώσεις μιας τέτοιας πρότασης. Αν δει κανείς την ομολογία της αποφάσης του, ΔΕ, του ε, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, την περίπτωση ΜΑΠΑ για παράδειγμα, επανειλημμένα και πάντα μπορούμε να το δούμε και να το πούμε ότι αυτά δεν ευθυγραμμίζονται σε σχέση με το άρθρο 7 και το άρθρο 8 της Σύμβασης για την προστασία της προσωπικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων και της οικογενειακής ζωής. Και γίνονται εξεταστικές έρευνες και διακριβώσεις έτσι εξεθρίασα και ε, συγκυριακά. Θα ήθελα να, πω, να αναφερθώ και στην οδηγία ε, καταχώρησης και αποθήκευσης ε, Retention Directive που απορρίφθηκε από συνταγματικά δικαστήρια όσον, των κρατών μελών όσον αφορά εκτελεστικές διατάξεις της ίδιας της οδηγίας. Υπάρχει ένα θέμα εκπροημίου σημαντικό που έχει οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό ε, συνταγματικό δικαστήριο και πρόκειται στο ΔΕΚ με συγχωρείτε και θα εξεταστεί και υπάρχουν σημαντικά σαφή θέματα επί όπως την ανάγκη να υπάρχει συνολική τέτοια αποθήκευση και καταχώρηση στοιχείων όσον αφορά την ανάγκη και αναγκαιότητα που απορρέει από μια δημοκρατική κοινωνία ή και στατιστικά στοιχεία που πρέπει να τηρούνται. Αν συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά με τα όσα συλλέγονται για τις, τους επιβάτες με έξι εξαμηνιαία περίοδο κατακράτησης το να αποθηκευτούν άλλα επί χρόνια και οι συνολικές σφαιρικές αναλύσεις όλων των δεδομένων επιβατών φαίνεται ότι δεν είναι λιγότερο επιθετική παρέμβαση αλλά περισσότερο παρεμβατική δράση. Θα έπρεπε να αναμείνουμε μια σαφή απόφαση του 10 προτού προχωρήσουμε παρακάτω και πάμε πιο πέρα στην έγκριση και υιοθέτηση αυτών των μέτρων. Επιπλέον θα ήθελα να πω ότι δεν βλέπω πολιτικά να είναι η σωστή οδός αυτή ώστε υπό το φως των συζητήσεων που είχαμε όσον αφορά την παρακολούθηση να συνεχίσουμε να έχουμε μέτρα παρακολούθηση σε ένα προληπτικό πλαίσιο. Πρέπει να έχουμε καλύτερη ανταλλαγή ε, στοιχείων όταν έχουμε θέματα επιβολής ε, του νόμου και δίωξης εγκλημάτων και συνεργασίας αρχών για την εξέταση και διακρύβωση εγκλημάτων και παραβάσεων ώστε να συλληφθούν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι εγκληματίες. Χρειάζεται βελτιωμένη συνεργασία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κοινέ προδιαγραφές κατά τα άλλα σίγουρα και συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων. Κοινέ προδιαγραφές για την ανταλλαγή πληροφοριών κοινέ τέτοιε προδιαγραφέ από την οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τη ΕΕ θα διασφαλιστεί. Αυτή πρέπει να είναι η βάση συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών για καλύτερη συνεργασία και σημαντικό βήμα για την καλύτερη ανταλλαγή στοιχείων και δεδομένων. Δεν βλέπω γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η οδηγία μπορούμε και ε, θα θέλαμε να έρθει επί και έτσι να εξεταστεί. Στο τέλος τέλος το τελευταίο επιχείρημα είναι να αντιμετωπιστούν τα θέματα της ε, γενικής ε, παρακολούθησης. Αυτά δεν είναι σύμβατα με τις αρχές κράτους δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ας εκπονήσουμε κοινέ προδιαγραφές για το τι θα ισχύει. Συμφωνώ να έχουμε μια κοινή συνάντηση, να συζητήσουμε την οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την Ευρωπόλ και την Υπηρεσία Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να συζητήσουμε τα σχετικά και μετά να δούμε ποια πορεία θα ακολουθήσουμε. Η κυρία Κόλτεμπαχ παρακαλώ. Ευχαριστώ θερμά. Σήμερα εκπροσωπώντας συνάδελφο θα ήθελα να τοποθετηθώ και εξ ονόματος της συναδέλφου να πω που παρακολύεται λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης να παραστεί για τη συζήτηση ε, στην Ευρώπη των θεμάτων PNR λόγω του ότι υπάρχουν σημαντικές επιφυλάξεις για την ανάγκη και αναγκαιότητα αυτών των μέτρων η σκοπιμότητα ενός τέτοιου μέτρου αμφισβητείται. Όλο και περισσότερη παρακολούθηση δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε βελτίωση της ασφάλειας. Περιστέλλεται η ελευθερία όμως, συρρυκνώνεται η ελευθερία και στο τέλος τέλος η καταπολέμηση τρομοκρατίας και εγκλημάτων δεν μπορεί να οδηγεί σε αυτήν την κατάσταση. Και για την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στο Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα επιχειρήματα, πολύ καλά με 30 ψήφους ε, κατά ε, απέρριψε αυτή την πρόταση. Δεν είναι αποδεκτό να, να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για παλαιές τροπολογίες που την προηγούμενη φορά, τελευταία φορά δεν εξετάστηκαν, ε, μια και η οδηγία απορρίφθηκε συνολικά. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς προς όφελος των πολιτών και υπέρ της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους, πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτή την απόρριψη και σε σχέση με τα όσα γίνονται από φιλικές χώρες με το πρίσμα και το τέμπορα συλλέγονται δεδομένα χωρίς καμιά άδεια αυτό δεν προάγει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κανείς δεν θα καταλάβαινε τώρα αν θα είχαμε μια τόσο σημαντική αλλαγή σε σχέση με την απόρριψη που ακολουθήσαμε πώς μπορούμε να την ανατρέψουμε. Ευχαριστώ. Ε, Εσείς στη συνέχεια παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ακολούθησα τη συζήτηση με ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Διότι πίστευα ότι είχε γίνει ήδη η ψηφοφορία. Έγινε αυτή η ψηφοφορία και είχαμε λοιπόν ε, την ε, ίδια αυτή απόφαση που είχε ληφθεί και δεν μπορούμε να την ανατρέψουμε. Μας αναφέρθηκε εδώ η απόρριψη, του συμβιβασμού. Αυτή ήταν νομίζω όμως και η πρόθεση ευθύς εξ αρχής και τώρα υπάρχει επιθυμία να καταλήξουμε σε νέες λέει διαπραγματεύσεις. Πρέπει να ρυθμιστούν τα πλαίσια σε σχέση με τα κράτη-μέλη βέβαια, αλλά αυτό δεν είναι και επιχείρημα από την άλλη πλευρά. Ασφάλεια και δικαιοσύνη είναι κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών μελών υπό τη συνθήκη. Και θα ήταν το χειρότερο αυτό το οποίο θα μπορούσε να συμβεί. Να έχουμε αποτέλεσμα το οποίο δεν θα προήγε την Ευρώπη, αλλά θα την ε, ε, αναχέτιζε. Είχαμε όμως μια ψηφοφορία που έγινε και ψηφίσαμε σχετικά. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι αυτό ήταν μια δοκιμαστική, μια προσπάθεια πειραματική. Ήταν ψηφοφορία που έγινε, το αποτέλεσμα είναι δεδομένο, πρέπει να προσέξουμε να μην ανατρέψουμε θέματα τα οποία έχουν ήδη αποφασιστεί με βάση ψηφοφορία που έγινε. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να αναμείνουμε, να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τα κράτη-μέλη, με τα δικαιώματα τα οποία έχουν υπό τους όρους της συνθήκης. Έχουμε εμείς δικαίωμα να επαναπέμψουμε θέματα στην Επιτροπή. Λοιπόν. Του έχω επανέλθω στον κύριο Κέκοπ. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα ήθελα να απευθύνουν κάποια σχόλια στην κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Επιτροπή Λίμπε, ναι ή όχι. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έλαβε γνώση της απόφασης της Ολομελίας την 10η Ιουνίου. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι συνεχίζεται η συζήτηση ε, στο Κοινοβούλιο για αυτήν την προτινόμενη οδηγία PNR που είναι μια σημαντική πρόταση. Σήμερα ακούσαμε με προσοχή όλες τις ανησυχίες που εγείρει η πρόταση αυτή και βεβαίως θα τις λάβουμε σοβαρά υπόψη. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες έτσι ώστε να εγκριθεί η οδηγία αυτή. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια και για τις εθνικές δραστηριότητες. Επανειλημμένα έχει πει η Επιτροπή απαντώντας και σε γραπτή ερώτηση 60 χώρες έχουν ε, ζητήσει χρημοδότηση σχετικά ε, με την παροχή τέτοιων πληροφοριών όπως αυτές που προβλέπονται από την ε, νομοθεσία. Πολλές ε, χώρες μέλη λαμβάνουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να δημιουργήσουν συστήματα PNR. Κατά την άποψη της Κομισιόν αυτό ε, εντείνει την άποψη ε, για την ανάγκη ύπαρξης ομοιογενούς προσέγγισης σε ενωσιακό επίπεδο. Λαμβάνουμε υπόψη μας τις λεπτομέρειες αυτών των δραστηριοτήτων και θα επανέλθουμε βεβαίως. Το Συμβούλιο, λέει ο Πρόεδρος, θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Όχι. Επομένως κύριε Κίρκοπ, ο εισηγητή μας λοιπόν, ο κύριος Κίρκοπ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, παρά κάποιε επιφυλάξει, πιστεύω ότι γενικώ η συζήτηση ήταν θετική. όμω να διευκρινίσω κάποια στοιχεία. Ένα προς τον κύριο Άλμπρεχτ. Ε, κύριε Άλμπρεχτ, είναι δημοκρατικών ε, αντιλήψεων και κατανοεί φαντάζομαι ότι δεν είναι αρκετό να πει κανείς ότι μια επιτροπή αποφάσισε κάτι, άρα το κοινοβούλιο ε, θα το στηρίξει. Από όσο ξέρω εγώ, οι διάφορες επιτροπές κάνουν προτάσεις τις οποίες υποβάλλουν στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Ε, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν λίγο τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, να δουν πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ε, είναι προς συμφέρον όλων να γνωρίζουμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα πράγματα. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της οδηγίας, βεβαίως είναι ε, πολύ περίπλοκο ζήτημα και ο κύριος Άλμπρεχτ και η κυρία Ίντβελτ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ε, και ενδεχομένως θα προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά ε, χρειάζεται κάποιος χρόνος η Κομισιόν και μόλις τώρα το ξαναείπε ότι έχουμε μια κατάσταση όπου ε, δημιουργούνται συστήματα PNR χωρίς προηγούμενη ε, συμφωνία. τα πρότυπα, τα στάνταρτ, ε, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις ε, τις οποίες ε, θα θέσουμε σε ένα σύστημα ευρωπαϊκό PNR θα πρέπει να εφαρμόζονται και από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δώσουμε αυτές τις βασικές αρχές και τα βασικά εχέγγυα όσον αφορά τις πληροφορίες κτλ. Θα πρέπει να υπάρξουν τυποποιημένες διαδικασίες που να ικανοποιούν και τις αεροπορικές εταιρείες που μεταφέρουν τους επιβάτες ε, και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα, μία σειρά προτύπων, όχι ένα κατακαιρματισμένο σύστημα, πολλά δηλαδή συστήματα στα οποία θα καταλήξουμε αν δεν έχουμε συμφωνία επί του Ευρωπαϊκού Συστήματος PNR διαδικασίες τώρα ε, και εμείς πιστεύουμε ότι διαδικαστικά πρέπει να προχωρήσουμε ε, με κατεπίγουσα διαδικασία. Θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, πρέπει να δώσουμε όλες τις, ε, να κάνουμε όλες τις συζητήσεις γρήγορα για τις οδηγίες. Πολλούς μήνες περιμένουμε. Ε, τα ζητήματα αυτά και τα συζητούμε. Θα, θα έχουμε και άλλη συζήτηση. Κυρία Ρομέρο Λόπες, είναι μια καλή ευκαιρία να ασχοληθούμε με τα ε, ακαθόδη ζητήματα και θα το κάνω εγώ σαν εισηγητής. Ελπίζω ότι τώρα θα προχωρήσουν τα πράγματα και διαβεβαιώνω τους συναδέλφους ότι θα είμαι ανοιχτός σε συνεργασία όσο περισσότερο μπορώ. Ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν. Τα τελικά σχόλια του εισηγητού τα ακούσαμε. Και επομένως θα συνεχιστεί η συζήτηση, εάν συμφωνείτε, να περάσουμε στο σημείο 7 που αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων πρέπει να έχουν θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και επίσης κατάλογο αυτών των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση. Η συγγήτρια είναι η συνάδελφος Μαρία Γκαμπριέλ. Σας βλέπω να είσαστε εδώ. Θα ακούσουμε λοιπόν τη γνώμη της εισηγητρίας και μετά θα ανοίξουμε τη συζήτηση έτσι ώστε και οι άλλοι συνάδελφοι και το Συμβούλιο και οι Κομισιόν να μπορέσουν να πάρουν το λόγο. Κυρία Γκαμπριέλ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους οικειώδης συγητής. Παρακαλώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, αυτοί που εγκαταλείπουν την αίθουσα, παρακαλώ να την εγκαταλείψουν ησύχως χωρίς να προκαλούν αναστάτωση στην αίθουσα. Κυρία Γκαμπριέλ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου για τον τακτικό και επικοδομητικό διάλογο που εξ αρχής ε, μας έδωσε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην εξέταση αυτού του φακέλου έχοντας πλήρη γνώση των στοιχείων. Ε, να σας θυμίσω ότι η 139 ε, του 2001 καθορίζει τον θετικό και τον αρνητικό κατάλογο. Χώρες, το κατάλογος των χωρών δηλαδή που χρειάζονται η υπηκοή τους θεώρηση και αντίστοιχα αυτοί που δεν χρειάζονται. Να πω πρώτα απ' όλα ότι εδώ η τροποποίηση είναι έκθεση παρακολούθησης. Επίσης, ο διαχωρισμός θετικής και αρνητικής λίστας γίνεται με ανάλυση αναπερίπτωση βάσει κριτηρίων που κυρίως συνδέονται στη λάθρομετανάστευση, ε, στη δημόσια ασφάλεια, στην ασφάλεια γενικότερα, στη δημόσια τάξη ε, και λαμβάνει υπόψη επίσης ε, δύο αρχές την περιφερειακή συνοχή ε, και την αμοιβαιότητα. Ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι εξελίσσονται οι δύο αυτές αρχές το χρόνο, ε, πρέπει σε τακτικά διαστήματα να αναθεωρούνται οι θετικές και αρνητικές λίστες. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θέλει να επικαιροποιήσει τον ε, κανονισμό αυτό η Κομισιόν. Στο αρχικό της κείμενο η Κομισιόν κάνει τρεις προτάσεις ε, βάσει τριών επεξηγήσεων. Ε, με τον ίδιο τρόπο θα διαρθρώσω και εγώ την παρουσίασή μου. Δηλαδή θα αναφερθώ στις αιτίες και μετά στα σχόλια που έχω σαν, και συστάσεις που έχω σαν εισηγήτρια. Πρώτον, η Κομισιόν λοιπόν ζητάει ε, για την ε, Δομινική Δημοκρατία, Μάρσαλ, Μικρονησία, Λαρούα, Παλάους, Αγία Λουκία, ε, Γρεναδίνη, Τιμόρ, Ανατολικό Τιμόρ, Τρινιδάδη Τομπάγκο κτλ. Προτείνει λοιπόν να μην χρειάζονται πλέον οι υπήκοοι αυτών των χωρών την θεώρηση. Αυτό σημαίνει ότι οι υπήκοοι ε, θα ε, ε, επιτύχουν αυτήν την αφαίρεση από τον ε, ε, κατάλογο με την υποχρέωση θεώρησης εφόσον υπογραφούν οι διμερείς συμφωνίες. Ε, δεύτερη πρόταση. Για όλους τους Βρετανούς υπηκόους που δεν, που δεν έχουν γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Βόρεια Ιρλανδία βάσει του δικαιώματος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κύριε Πρόεδρος, παρακαλώ πολύ να μην φωνασκούν τα, οι Αυτή τη στιγμή ένας βουλευτής ομιλεί και παρακαλώ πολύ να την σεβαστείτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τρίτη πρόταση αφορά την αρνητική λίστα. Η Κομισιόν προτείνει τον Νότιο Σουδάν να περιληφθεί στον κατάλογο των χωρών οι υπήκοοι των οποίων ε, ε, ε, υποχρεούνται να έχουν βίζα, θεώρηση για τη διέλευση εξωτερικών συνόρων. λοιπόν, τώρα να αναφερθώ στις επεξηγήσεις οι οποίες δικαιολογούν ε, τις ε, δύο πρώτες ε, κατηγορίες οι οποίες απαλλάσσονται από την υποθεώρηση βίζας. Θεώρηση. Όσον αφορά της, τα νησιά του Ειρηνικού και της Καραϊβικής. Οι χώρες αυτές δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο όσον αφορά τα τρία ζητήματα τα οποία αναφέραμε στην αρχή. Και ως εισηγήτρια Θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξω την ε, μετάθεση των χωρών στη θετική λίστα, ε, διότι οι πολίτες τους αντιμετωπίζουν διπλό ε, βάρος, δηλαδή θα πρέπει να ζητήσουν και επιπλέον θεώρηση για τις χώρες Σέγγεν, άρα και μεγάλο οικονομικό βάρος. Ε, όσον αφορά τις, ε, τα έγγραφα ταξιδίου τα οποία δίνουν αυτές οι τρίτες χώρες δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως μπορούμε ε, να πούμε ότι ούτως ή άλλως τα, η ύπαρξη βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια αποτέλεσε το σημείο καμπής για τις χώρες των Ανατολικών Βαλκανίων έτσι ώστε να μπουν στο θετικό κατάλογο επομένως και για τους υπηκόους τη της ε, ε, Αγίας Λουκίας, Τρινιδάδη τον Πάγκο κλπ. έχουν ήδη ε, τα διαβατήριά τους τέτοια βιομετρικά χαρακτηριστικά, μπορούν να αναγνωστούν από τα ειδικά μηχανήματα και οι υπόλοιπες χώρες σύντομα πρόκειται να το πράξουν. Δεύτερον, ε, η ειδική κατηγορία των Βρετανών υπηκών. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η ομάδα που αναφέρεται στο σημείο 3 του παραρτήματος 1 δεν παρουσιάζουν πρόβλημα όσον αφορά την λαθρομετανάστευση προς τον χώρο Σέγγεν και ότι οι περισσότεροι μεταξύ αυτών ζουν στις ε, ε, νήσους της Καραϊβικής ε, και έχουν ε, μια καλή σχέση και με τις ε, υπόλοιπες γειτονικές χώρες οι οποίες, το των οποίων δεν έχουν υποχρέωση θεώρησης η ενημέρωση τώρα της αρνητικής λίστας με τη συμπερίληψη του Νοτίου Σουδάν. Να υπενθυμίσω ότι την 9 Ιουλίου του 2011 επισήμως έγινε ανεξάρτητη χώρα το Νότιο Σουδάν σε σχέση με το Βόρειο Σουδάν το παράρτημα 1 λοιπόν θα πρέπει να ε, τροποποιηθεί δεόντως αναφερόμενο στις νέες χώρες του κόσμου. Όσον αφορά τις ε, τρεις κατηγορίες που ανέφερα προηγουμένως, ε, μπορώ να πω ότι συμφωνώ με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ως εισηγήτρια θέλω να κάνω κάποιες άλλες συστάσεις. Πρώτον, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την υποχρέωση ε, θεώρησης ε, για τα μέλη της Ισομερούς ε, Συνέλευσης ΑΚΕΟΚ όταν ταξιδεύουν για να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις της Ισομερούς Συνελεύσεως. Δεύτερον, εκφράζω έντονη επιθυμία ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί πλήρως και σε πραγματικό χρόνο να πληροφορείται για το καθεστώς των διμερών συνθήκων και την ε, ε, όποια εφαρμογή αυτών των συνθήκων. Δηλαδή θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρομαι στην υποχρέωση σεβασμού του δικαιώματος πληροφόρησης που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε, όλες, σε όλα τα στάδια ε, και εν πάση περιπτώσει ένα εξάμενο. Επίσης καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, πληροφορεί άμεσα το Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε πληροφόρηση ε, ε, λαμβάνει και η οποία αφαιρεί την ανέρεση κάποιας συμφωνίας. Όσον αφορά τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στην παρούσα πρόταση σε αιτιολογική σκέψη. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του κανονισμού έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στο διατακτικό σε κάποιο άρθρο ε, αυτό το περιεχόμενο της ιδεολογικής σκέψης. Τέλος, όσον αφορά τα παραρτήματα και τον τρόπο με τον οποίο και οφείλουν να ενημερώνονται, Επιμένω ότι αυτό είναι ένα σημείο αναφοράς. Πρέπει να ξέρουμε οποιαδήποτε ε, χρονική στιγμή με ποιο τρόπο τροποποιούνται ή ενημερώνονται αυτά τα ε, παραρτήματα και κατά αυτήν την έννοια θα ήθελα ε, να υπάρξει ε, σκέψη σε βάθος έτσι ώστε να δούμε μήπως ε, σύμφωνα με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να, μάλλον μήπως πρέπει να διέπονται από κατεξουσιοδότηση πράξεις αυτές οι επικαιροποιήσεις. Αυτά ήθελα να σας πω. Παραμένω βεβαίως ανοιχτή σε οποιαδήποτε συζήτηση, πρόταση, σύσταση, σχόλιο, παρατήρηση των συναδέλφων, τους οποίους εκ των προτέρων ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γκαμπριέλ. Κυρία Ιντβελτ. Uh, Ευχαριστώ. Θα αναγνώσω μια δήλωση του σκιο... της σκιώδους η οποία δεν μπορεί να είναι εδώ. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της στα γαλλικά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετικό έργο της καθώς επίσης και για την συνεισφορά των σκιωδών. Συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής να καταργηθεί η υποχρέωση θεώρησης. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα προς τις ε, χώρες εκείνες, καθώς επίσης διευκολύνει και τις επαφές με τους υπηκόους αυτών των χωρών. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με βάση τις μεταναστευτικές ροές και τη σχέση με αυτές τις χώρες. η κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης έχει πολλές ε, επιπτώσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, όπως ε, για παράδειγμα η αύξηση του αριθμού των τουριστών από τις χώρες αυτές. Οι προτινόμενες αλλαγές αναφέρονται σε χώρες οι οποίες δεν, δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα, κανένα κίνδυνο μετανάστευσης ή ε, δημόσιας τάξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρομαι στις χώρες ΑΚΕ. Στις ισομερείς στην, ισο... μάλλον στην ισομερή συνάντηση ε, με τις χώρες ΑΚΕ τον Άγιο Δομήνικο τον Φεβρουάριο πολλοί εκπρόσωποι αντιμετώπισαν προβλήματα γιατί ε, χρειαζόντουσαν ε, θεωρήσεις για να παρευρεθούν. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να δώσουν ε, εξαιρέσεις, να παραχωρήσουν εξαιρέσεις από αυτή την υποχρέωση θεώρησης για τα μέλη της ισομερούς συνέλευσης ΑΚΕ, καθώς ε, επίσης και για τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την περιοχή. Τα θέματα αυτά τα συζητήσαμε και με τους σκιώδους εισηγητές και στην έκθεσή της η κυρία Γκαμπριέλ ζητά να επαναξεταστεί λοιπόν το ζήτημα για εκείνους που προέρχονται από τις χώρες ΑΚΕ και συμμετέχουν στις συναντήσεις εκτός, σε χώρες εκτός Σέγγεν και συμφωνώ πλήρως με αυτή την πρόταση της κυρίας Γκαμπριέλ. Θα βοηθήσει να υπάρξει σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΑΚΕ. Την έκθεση που υιοθετήθηκε στην Σύνοδο και Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 είχε αναφερθεί η δυνατότητα να εξεταστεί το ζήτημα παραχώρησης θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων σε εκείνους που ταξιδεύουν συχνά και προέρχονται από τις χώρες ΑΚΕ. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν που έχει συζητηθεί στην, ε, στην μερίς με τις χώρες ΑΚΕ και θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της αμοιβαιότητας. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να υιοθετήσει, να εφαρμόσουν μάλλον τις συστάσεις τις οποίες υιοθέτησε η Συνέλευση ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ε, δεσμεύομαι από την πλευρά μου να το κάνω ε, προς το Βέλγιο, δεδομένου ότι σε πολλές συναντήσεις που διοργανώνονται στο Βέλγιο εκπροσωπούνται άτομα από τις χώρες ΑΚΕ. Ακούσαμε λοιπόν τη ε, κυρία Σκηνή και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Έντσιου. Μαρία, να σας συγχαρώ για την παρουσίασή σας και ε, εκ μέρους της κοιόδους της ηγετρίας των Σοσιαλδημοκρατών που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα θα σας μεταφέρω την άποψή της. Η Τάνια λοιπόν είχε μια πολύ καλή συνεργασία μαζί σας την οποία εκτιμά και θεωρεί ότι ήταν πολύ επικοδομητική. Σας ευχαριστώ για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει πάνω σε αυτό το φάκελο και υποστηρίζει την εκθεσή σας η Τάνια. Καλωσορίζει την πρόταση της Επιτροπής ως έχει. Τη θεωρεί εξαιρετικά ισορροπημένη και υποκοδομητική. Επίσης καλωσορίζει το προσχέδιο της έκθεσης που έχετε ετοιμάσει. Ε, θεωρεί ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και προσβλέπει στην μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχουν τη δυνατότητα η Επιτροπή και το Συμβούλιο να, μιλήσουν. Ο ε, κύριος Πάλμαν, ε, εκπρόσωπος της Επιτροπής, πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και σε όλους. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την ε, έκθεση, την οποία προφανώς καλωσορίζουμε γιατί καταρχήν είναι ε, υπέρ της ε, θέσης της Επιτροπής. Ε, επίσης όμως η εισηγήτρια κάνει διάφορες συστάσεις και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές πιο λεπτομεριακά. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια σύσταση προς την Επιτροπή να ενημερώνει, να, να φροντίζει το Κοινοβούλιο να γνωρίζει διαρκώ πώ εξελίσσονται διαπραγματεύσεις, ε, οι διμερεί διαπραγματεύσει για τι σχέσει με τι θεωρήσει. Φυσικά, εμεί πάντα ε, επιθυμούμε να είναι πλήρω ενήμερο το Κοινοβούλιο για την εξέλιξη αυτών των διαπραγματεύσεων και οποιοδήποτε άλλου συναφού ζητήματο. Το ίδιο ισχύει και για διμερείς συμφωνίε άρσης τη υποχρέωση θεωρήσεων. παρόλο που δεν προβλέπεται θεσμικά μια τέτοια ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Από την δικιά μας την πλευρά ε, δεσμευόμαστε ότι θα του ενημερώνουμε οποτεδήποτε προβλέπεται η λήψη μια της τέτοιας απόφασης. Τώρα σε σχέση με την πρόταση να εισαχθεί στο διατακτικό σε κάποιο άρθρο ε, το κατάλογος των κριτηρίων για την άρση των θεωρήσεων είναι ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση και θα τη σκεφτούμε. Όμως εκ πρώτης όψεως νομίζω ότι τα κριτήρια, του γεγονός μάλλον, τα κριτήρια αυτή τη στιγμή ε, βρίσκονται στις αιτιολογικές σκέψεις, δίνει μια μεγαλύτερη ευελιξία στην Επιτροπή ε, όταν εξετάζει ποια χώρα, για ποια χώρα μπορεί να αρθεί η υποχρέωση θεώρησης. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφθήνει τον προηγούμενο Νοέμβριο, περασμένο Νοέμβριο, μια ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, στην οποία αναφέρεται ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις του παραρτήματος 139 θα λαμβάνουμε υπόψη μας και άλλα κριτήρια, κυρίως εκείνα που αναφέρονται στον οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει μια τέτοια άρση της θεώρησης. Με αυτό το σκεπτικό νομίζω είναι ενδιαφέρουσα η πρότασή σας, αλλά πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο. Τώρα σε σχέση με τα μέλη της ε, συνέλευσης ΑΚΕ που το έθιξε ε, και η κυρία Ιντφέλτ, εκ του κυρίου Μισελ, γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει αυτά τα μέλη της συνέλευσης ΑΚΕ και έτσι στο πλαίσιο της συζήτησης ε, για την μετανάστευση που έχουμε μαζί με τις χώρες ΑΚΕ έχουν ήδη εφετηθεί δύο συστάσεις. Τις ανέφερε η κυρία Ινφέλτ. Ξεκινήσαμε λοιπόν να επεξεργαζόμαστε τον τρόπο εφαρμογής αυτών των συστάσεων. Επικοινωνήσαμε ε, με τις βελγικές αρχές και τους υποβάλαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρώτη να αναθεωρήσουν ε, τον κώδικα θεωρήσεων έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα παροχής θεωρήσεων ε, πολλαπλής εισόδου πρώτον και δεύτερον να επιταχυνθούν οι διαδικασίες παροχής θεωρήσεων για τα μέλη εκείνα της συνέλευσης ΑΚΕ. Προτείνουμε λοιπόν η κάθε χώρα ΑΚΕ να καταρτήσει έναν κατάλογο με τα μέλη ε, της χώρας αυτής που συμμετέχουν στη συνέλευση, να την αποστείλει στην γραμματεία της συνέλευσης ΑΚΕ, η οποία θα τις ε, ε, συμπτύξει όλες μαζί και μετά η γραμματεία θα προωθήσει αυτόν τον κοινό κατάλογο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θα τον αποστείλουμε τον κατάλογο στις βελγικές αρχές, οι οποίες μετά θα ε, τον αποστείλουν στις βελγικές ξενικές αρχές της χώρας και αναφερόμαστε στο Βέλγιο εδώ ε, έτσι ώστε ε, οι βελγικές αρχές να γνωρίζουν, να γνωρίζουν ποια είναι τα μόνιμα μέλη που συμμετέχουν σε αυτές τις συναντήσεις και όταν αυτά τα μέλη λοιπόν κάνουν αίτηση για μακράς διάρκειας θεώρηση να τους παρέχετε γρήγορα. Μια ακόμα πρόταση αφορά τις επιτεχημένες διαδικασίες. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί ότι θα αποστείλει όσο το δυνατόν γρηγορότερα μέσω από τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής στις χώρες αυτές έναν κατάλογο στις τοπικές αρχές που θα έχει τις ημερομηνίες διαξαγωγής συναντήσεων στο πλαίσιο του διαλόγου ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημαίνει ότι και τα βελγικά προξενικά προξενία θα γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι ημερομηνίες και θα μπορούν να διευκολύνουν τους, ε, τα μέλη των συναντήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανταποκρίνονται στα αιτήματα τους για θεώρηση πολύ πιο γρήγορα. Αυτό λοιπόν το σύστημα έχουμε ξεκινήσει να δημιουργούμε. Προφανώς υπάρχει αμοιβαιότητα εδώ, δηλαδή από την πλευρά τους οι χώρες ΑΚΕ θα πρέπει και εκείνες να διασφαλίσουν ότι δεν θα περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή τα μέλη ε, της Συνέλευσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλουν το αίτημα θεώρησης όπως δυστυχώς πολύ συχνά συμβαίνει. Θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα τους εγκαίρως για να έχουν και την απάντηση εγκαίρως. Τέλος, προτείνεται να σκεφτούμε την χρήση πράξεων κατά εξουσιοδότηση για την επικαιροποίηση του καταλόγου. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί συχνά με τη χρήση ε, πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν σκόπιμο σε αυτήν την περίπτωση, γιατί μιλάμε για ενημέρωση ενός κατάλογου, καταλόγου, ο οποίος όμως είναι η ουσία της οδηγίας 159 και νομίζω ότι δεν ε, επιτρέπεται και με βάση τη συνθήκη να μεταβάλλεται η ουσία μιας ε, οδηγίας με βάση ενός κανονισμού μάλλον με βάση κατεξουσιοδότησης εμπράξης. Με τη διαδικασία της ε, συναπόφασης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί ε, τις αρμοδιότητές του και έχει πολύ μεγαλύτερο λόγο σε σχέση με εκείνον που θα είχε αν η Επιτροπή χρησιμοποιούσε κατεξοσιοδότηση πράξης. Πάντως θα το εξετάσουμε συμπερασματικά να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για το, την θετική σας έκθεση και βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Το Συμβούλιο. Θέλετε κι εσείς. Ναι. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και εμείς την εισηγήτρια για την έκθεση καλωσορίζουμε την πλειονότητα των συστάσεών της. Διαφωνούμε όμως με την τελευταία ε, πρότασή της, μιας και πρόκειται για ε, φάκελος συναπόφασης. Εμείς δεν θεωρούμε ότι οι κατεξουσιοδιώτες πράξη είναι σκόπιμες ή ε, ο ενδεδειγμένος τρόπος. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε με τις προτάσεις της εισηγήτριας, το Συμβούλιο προτινόμενες αλλαγές στον κατάλογο, θα θέλαμε επίσης να καταγραφεί, αν και σημειώνουμε την παρατήρηση της κυρίας Γκαμπριέλ για την περιφερειακή συνοχή, πρέπει να, να σημειώσουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός κρατών του Συμβουλίου προτείνει να συμπεριληφθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε αυτόν τον κατάλογο. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επ' αυτού πριν να λάβουμε την τελική μας απόφαση. Αυτά ήταν τα κύρια σχόλια που ήθελα να κάνω για την έκθεση και να επισημάνω ότι η συνεργασία μεταξύ της Ιγήτριας και της Ιρλανδικής Προεδρίας ήταν εξαιρετική. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και ευελπιστούμε ότι τέτοια καλή συνεργασία θα έχουμε και υπό τη Λουθουανική Προεδρία. Για να, ευελπιστώντας ότι θα καταφέρουμε να κλείσουμε το φάκελο σύντομα. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Καπριέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους κοιόδης που με στήριξαν και εκφράστηκαν θετικά υπέρ της ε, προτάσεώς μου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί μας έδωσε λεπτομερείς απαντήσεις όσον αφορά τις διάφορες συστάσεις που γίνονται στο κείμενο. Ε, θα ήθελα να πω σε σχέση με την τελευταία παρατήρηση για τα του Συμβουλίου για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως είπατε είναι μια πρόταση η οποία έφτασε αργά ε, και επομένως δεν συμπεριλαμβανόταν στην αρχική πρόταση της ε, Κομισιόν. Και εγώ δεν ετόλμησα ε, να αναφερθώ σε αυτό το θέμα ως εκπρόσωπος εισηγήτρια του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, 11 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Βάσει των τροπολογιών θα συζητήσουμε έτσι ώστε το Κοινοβούλιο ε, να εκφραστεί υπέρ ή κατά των διαφόρων προτάσεων που γίνονται στην έκθεση. Για μία ακόμα φορά ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετικά καρποφόρα συνεργασία με όλους τους χειώδεις ηγητές. Πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε αυτόν τον τακτικό και επικοδομητικό διάλογο θα καταφέρουμε ε, σε έφετο χρόνο να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό στέλνοντα το μήνυμα και ε, σε όλες τις χώρες οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι η 11η Ιουλίου έχει οριστεί ε, ε, το μεσημέρι, 12η μεσημβρινή, έχει οριστεί ως προθεσμία υποβολής των τροπολογιών. Έχουμε τώρα το σημείο 8, το οποίο αφορά την ίση μεταχείριση προσώπων εξαιτούς της που πεπιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετησίου προσανατολισμού. Είναι, αναφέρεται στη λεγόμενη οριζόντια ε, οδηγία για την έλλειψη διακρίσεων. Ήρεμα παρακαλώ όλοι, όχι πηγαδάκια, όχι συζητήσεις μέσα στην αίθουσα. Όσοι εγκαταλείπουν την αίθουσα να το πράξουν ησύχως παρακαλώ. Έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Please. Ε, Σας έλεγα ότι αυτό το σημείο, δηλαδή αυτή η οριζόντια ε, οδηγία μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και πριν ξεκινήσει αυτή η θητεία είχε αρχίσει να εμφανίζεται κατά διαστήματα το θέμα αυτό. Το 2008 ξεκίνησε η μακρά πορεία και ακόμα δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή την οριζόντια οδηγία. Έχει για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα μπλοκαριστεί το θέμα στο Συμβούλιο, γιατί εκεί χρειάζεται, ε, χρειάζεται ομοφωνία για το θέμα αυτό. Ξεκίνησε πάντως να, μας να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό στην ε, λεγόμενη έκθεση Μπρούκεμπρεκ το 2009, Σεπτέμβρη. Και τώρα, μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης ε, της ε, Λισαβόνας, το θέμα ε, βασίζεται στο άρθρο 19 της συνθήκης λειτουργίας. Επομένως, ζητείται η συνένεση του Κοινοβουλίου. Είναι βάση της διαδικασίας συνενέσεως αυτή. Ε, η έκθεσή του, αλλά θέλουμε ακριβώς να ακούσουμε από την Ιρλανδική Προεδρία, από το Συμβούλιο δηλαδή, τα νέα. Να μας πούνε αν έχει γίνει καμία πρόοδος, πού βρισκόμαστε τέλος πάντων όσον αφορά το θέμα αυτό. Να ακούσουμε πρώτα τι έχει να μας πει ε, η Ιρλανδική Προεδρία και μετά να μας πει ο εισηγητής μας, ε, κύριος Ρωμέδα, τι γίνεται. Brian, ναι. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, η πρόταση αυτή προχωράει με πολύ αργό ρυθμό. Όπως σας έλεγα λοιπόν, η πρόταση αυτή προχωράει με πολύ αργό ρυθμό. Δεν είμαι σε θέση και δεν επιτρέπεται να σας πω ποια είναι η θέση των μεμονωμένων μερών, αλλά δεν σας ε, κομίζω γλάφκα εάν ε, σας πω ότι κάποιες χώρες ε, δεν συμφωνούν. Υπάρχει μια μεγάλη, ένα μεγαλύτερο βέβαια μέρος χωρών, αριθμός χωρών ε, που συμφωνούν, στηρίζουν την πρόταση της Κομισιόν. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αμφιβολίες στον αφορά το κείμενο και προσπαθούμε να τις λιάνουμε. στην Ιρλανδία έχουμε ε, εξ αρχής ε, δηλώσει ότι έχουμε μια θετική εμπειρία όσον αφορά ε, την διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και ατόμων και θέλαμε να μεταφέρουμε την εμπειρία μας εδώ. Πάντως πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία νέα αρχή, δεν υπάρχει τίποτα καινούριο ε, στο κείμενο που να μην υπάρχει ήδη και να μην προβλέπεται από την ε, εσωτερική Ιρλανδική νομοθεσία. Πρέπει να πω ότι ε, υπάρχουν περισσότερες αναφορές σε διευκρινήσεις και ελέγχου στην εσωτερική μας εθνική νομοθεσία. Υπό το φως αυτό ο στόχος που είχαμε θέσει στην ε, Ιρλανδική Προεδρία ήταν να λιάνουμε όσο γίνεται περισσότερα από τα στοιχεία, ε, να ε, διασκεδάσουμε τις περισσότερες από τις ανησυχίες και επομένως να οδηγήσουμε το Συμβούλιο να λάβει μια πολιτική απόφαση επί της αρχής. Εστιαστήκαμε κυρίως σε μια σειρά ζητημάτων στην, τα οποία αναφέρονται στην έκθεση πρόοδου, πρόοδου, όπως ας πούμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση σε στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ε, ασφάλιση. Πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία σημαίνει ότι ε, αυτές, ε, η οργάνωση αυτών των στοιχείων θα είναι εθνική αρμοδιότητα. Επίσης η δημιουργία υποδομών για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία επίσης ε, την, ε, το, το σημείο της, ε, του γενετήσου προσανατολισμού, αυτό δηλαδή να μην αποτελεί σε καμία περίπτωση αιτία διακριτικής μεταχείρισης. Επίσης να μην υπάρξει καμία διαφορετική τιμολόγηση βάσει όλων αυτών των ιδιαιτεροτήτων των ομάδων που αναφέρουμε όσον αφορά την τιμολόγηση παροχής υπηρεσιών. Ε, επίσης, βάσει της αξιολόγησης αντικτύπου της εσωτερικής μας νομοθεσίας τα τελευταία 13 χρόνια, μπορώ να πω ότι ε, δεν ε, θα ε, υπάρξει βάση της νέας προκεινόμενης νομοθεσίας οποιαδήποτε αύξηση του βάρους διοικητικού άκτους λοιπά για τις νέες χώρες. Εν πάση περιπτώσει προβλέπουμε και μία νέα πράξη, την πράξη για την βελτίωση της προσβασιμότητας όπου θα αναφέρονται ακριβώς πιο ιδιαίτερα στοιχεία. Ε, η έκθεση πρόοδου θα πρέπει να προχωρήσει ε, και οι πρόνοιες ε, οι οποίες αναφέρονται σε χρηματοδοτικές υπηρεσίες και κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να τύχουν λεπτομερούς και εξετάσεως. Η Λιθανική Προεδρία ε, όχι μόνο θα συνεχίσει να μελετά το κείμενο, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει να το μελετά και ενδεχομένως ε, το κείμενο να είναι έτοιμο σε λίγο για την πολιτική απόφαση την οποία να ανέφερα προηγουμένως. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας. Ο εισηγητής μας τώρα να πάρει το λόγο. Όχι, η Κομισιόν πρώτα. Ωραία, θέλει η Κομισιόν να πάρει το λόγο. Ο κύριο Σίβεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους σας. Εξ ονόματο τη Επιτροπή, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Ιρλανδική Προεδρία για την προσπάθεια την οποία κατέβαλε και την σημαντική εργασία την οποία έχει ήδη ε, κάνει όσον αφορά ε, το θέμα αυτό. Προχωρήσαμε πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες ε, ε, προεδρίες. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε ένα από τα σημεία τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Για πρώτη φορά έχουμε συνολικό ορισμό της έννοιας πρόσβαση, access. Ε, που ξεχωρίζεται πλέον ε, καθαρά από την επιλεξιμότητα όσον αφορά την εκπαίδευση κτλ. Λοιπόν, πρόσβαση σε κοινωνική προστασία, ε, σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, παιδείας, όσον αφορά την πρόσβαση σε υλικά αγαθά, υπηρεσίες κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε από την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών τα θέματα υγείας και ε, κοινωνικής ασφάλισης. Σε τεχνικό επίπεδο έχουν γίνει πρόοδοι, αλλά δεν έχει αλλάξει ακόμα η πολιτική κατάσταση. Είναι ίδια όπως την είχαμε γνωρίσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες εξακολουθούν για λόγους αρχής να αντιτίθενται στην οδηγία. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες αντιτίθενται σε συγκεκριμένες διατάξεις πρόνοιας δεν έχουμε ακόμα πολιτική ε, συμφωνία και επομένως ε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πάντως θα πρέπει να συνεχίσουμε με λογική και με ε, υπομονή και επιμονή να προλιάνουμε το έδαφος έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για την έγκριση όταν θα ανοίξει ένα παράθυρο πολιτικής ευκαιρίας. Δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί, ευελπιστούμε ότι θα συμβεί αρκετά γρήγορα. Εμείς έχουμε την πρόταση που υποβάλαμε πριν από πέντε χρόνια, εξακολουθούμε να τη στηρίζουμε. Ε, θα συνεργαστούμε με την Λιθουανική Προεδρία, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αναλάβει, θα λάβει την ε, σκητάλη από την ε, Ιρλανδική Προεδρία για το θέμα αυτό. Τώρα όμως ήρθε η ώρα του εισηγητού, ο κύριος Ρομέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και την Ιρλανδική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρώτο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω εδώ είναι δεν πρόκειται να επινοήσω να ανακαλύψω βέβαια κάτι καινούριο. Αλλά σε σχέση με την απογοήτευση είναι η πέμπτη το αφορά που έχουμε αυτή τη συζήτηση και δεν σημειώνεται καμία κίνηση. Δεν προοδεύουμε. Εξακολουθούμε να έχουμε τις ίδιες συζητήσεις όπως πριν από πέντε χρόνια και αυτό μας απογοητεύει, είναι πολύ απογοητευτικό. Για αυτή την πτυχή θέλω να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα μιας έννοιας ε, ενός θέματος που είναι σημαντικό για την προεκλογική περίοδο για την ε, προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές για την Ευρωβουλή του 2014 είναι η διαφάνεια, transparent. Αυτό είναι εκπληκτικό. Κάθε φορά ευθύνεται λέει ο πληθυσμός, ε, ε, ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δεν γίνεται κάτι. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν κινητοποιείται. Είναι κάποια πρωτεύουσα, κάποιες κυβερνήσεις κάποιων κρατών μελών που τροχοπεδούν τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι σε σχέση με τη διαφάνεια πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες μας και να ακουστεί δημόσια ποιος τροχοπεδεί τα πράγματα. Ο εισηγητής αυτός προς το Συμβούλιο ασκούσε πίεση για να προχωρήσουμε από τότε που αναλήφθηκε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δημόσια τοποθέτηση επ' αυτού γνωρίζουμε από εσωτερικές συζητήσεις, από προσωπικές επαφές διμερώς σε διάφορα επίπεδα, όλα αυτά τα πέντε χρόνια γνωρίζουμε ότι υπάρχει συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν προβλήματα. Είναι όμως πάρα πολύ ανησυχητικό για το, το ότι είναι τόσο δύσκολο να ονοματίσουμε, να κατονομάσουμε εκείνους που τροχοπεδούν αυτή τη συζήτηση και την οδηγούν στο να αποφευθεί να διεξαχθεί σε ένα δημόσιο πλαίσιο. Αυτό θέλω να αναφέρω εδώ και να το τονίσω. Δεύτερον, μας εκπλήσει επίσης ότι όλες οι τεχνικές πτυχές είναι τόσο δύσκολο να επιληθούν ουσιαστικά, όταν οι περισσότερες από τις χώρες που τροχοπεδούν αυτά τα πράγματα, οι ίδιες, οι ίδιες εσωτερικά αυτές οι χώρες στα νομοθετικά τους πλαίσια έχουν διασφαλίσει τις ουσιοδέστερες διατάξεις αυτής της ε, οδηγίας. Τα ίδια αυτά τα κράτη. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιος λόγος τεχνικά που να δικαιολογούσε την τροχοπέδηση χρόνο μετά χρόνο αυτών των θεμάτων από αυτά τα κράτη. Και είναι λοιπόν εδώ θα, ε, ε, μπορέσει, θα, θα σημειωθεί έκπληξη όταν διαπιστωθεί ότι συμβαίνει αυτό και ότι είναι τόσο δύσκολο παρόλα αυτά να βρεθούν λύσεις ε, όπως ε, για τεχνικά θέματα. Δεν αρνούμε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση. Όμως ε, τα δίθεν τεχνικά προβλήματα όπως αναφέρεται που δεν μπορούν να επιληθούν είναι πολύ εύκολο να επιληθούν αν θα υπήρχε πολιτική βούληση για να γίνει αυτό. Αυτό ζητάμε να γίνει και αυτό αναμένουμε από τις διάφορες προεδρίες. Το τρίτο σχόλιο που θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι. Εγώ δεν κατηγορώ όλες τις προεδρίες εξίσου. Το αναφέρω αυτό. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με διαφορετικές προεδρίες επ' αυτού. Κάποιες ήταν πιο επικοδομητικές, κάποιες λιγότερο επικοδομητικές. Ωστόσο πρέπει να ομολογήσω ότι σε προσωπικό επίπεδο με τους υπεύθυνους, ας τους αποκαλέσουμε έτσι, για την προαγωγή του χαρτοφυλακίου. Είχα προσωπικά καλές επαφές μέχρι τούδε. Το μόνο για το οποίο εκφράζω τη θλίψη μου εδώ είναι ότι είχα ζητήσει να συμμετάσχω ως εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου σε αυτές τις συζητήσεις για να ακριβώς μπορώ να συμμετέχω σε αυτές τις διαδικασίες. Ε, λοιπόν πρέπει να παραδεχθώ εδώ ότι δεν πέτυχα σε αυτό το αίτημά μου. Δεν στέφθηκε με επιτυχία. Κάποιες φορές μπόρεσε να γίνει δεκτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο από το Συμβούλιο να γίνεται δεκτό το αίτημα να διασφαλίζεται η ρήτρα ότι θα συμμετέχει το Ευρωκοινοβούλιο σε τέτοιες συζητήσεις. Διότι αυτό θα βοηθούσε στο τέλος τέλος στην προαγωγή αυτής της υπόθεσης. Αν θα υπήρχε ένα τέτοιο παράθυρο ευκαιρίας για να μπορούσε να ληφθεί μια απόφαση για αυτό το θέμα. Ίσως είμαι εγώ εκείνος ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι δυνατόν να μπορέσω να το καταφέρω κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας, όποιος και αν είναι, είναι σημαντικό να συμμετέχει με το Συμβούλιο σε αυτή τη διεργασία από πλευράς του Ευρωκοινοβουλίου. Να είναι σαφές λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διεργασίας ε, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει κίνδυνος ε, δίχασης ε, ε, κατακαιρματισμού αυτής της οδηγίας υπάρχουν κάποιες τάσεις ε, για να υπάρξει ένας διαχωρισμός, διαχωρισμός ε, σε σχέση με τα θέματα αυτά. Πράγμα το οποίο είναι απόλυτα επικίνδυνο. Και πάλι για άλλη μια φορά είμαι κάθετα αντίθετος στο να γίνει κάτι τέτοιο. Και στην έκθεση Μπότεμπεργκ είχαμε πει ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό για το Ευρωκοινοβούλιο. Παραμένω και εμένα σε αυτή τη θέση για το Ευρωκοινοβούλιο εγώ ως εισηγητής. Και επιμένω, όταν κάνουμε λόγο για αυτά τα θέματα δεν μπορούμε να ε, διχάσουμε ταυτότητες και να ξεχωρίσουμε ε, τέτοιου είδους θέματα επειδή θέλουμε να ευχαριστήσουμε μια κυβέρνηση ή μια άλλη. Αυτό είναι η γραμμή αφετηρίας, η γραμμή κίνησης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Είναι δεδομένη και ευελπιστώ ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα επιμείνει και θα εμείνει σε αυτή τη θέση και το ίδιο. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος κίνδυνος να γίνει τώρα κάτι τέτοιο, αλλά θέλω να το τονίσω αυτό, ότι είναι σημαντικό να μείνει αυτό συνολικά σε ένα πλαίσιο και να καλύψει όλα τα θέματα. Ας είναι λοιπόν σαφέ ότι μόνο στο, χώρο εργασίας μπορεί να διασφαλιστεί ε, η πτυχή της ποιότητας. Κι όμως δεν μπορώ να κατανοήσω πώς δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί αυτό σε όλες τις πτυχές ε, της καθημερινής ζωής. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να επεξηγήσω στους όσους εμπλέκονται. Είναι πολύ δύσκολο όμως να το αναγνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν γιατί. Γιατί υπάρχει μια τέτοια αναγκαιότητα υπό το ευρωπαϊκό πλαίσιο και δεν έχει διασφαλιστεί ακόμα. Και τέλος η τελευταία μου παρατήρηση. Ας κάνουμε λόγο για τη δημοκρατία λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι έκανε. Ζήτησε τουλάχιστον 12 φορές, 12 φορές ήδη οι εκπρόσωποι, οι εκπρόσωποι της, ε, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωβουλευτές, ε, ζήτησαν 12 φορές από το Συμβούλιο να απελευθερώσει αυτό το θέμα, να, να το αποτροχοπεδίσει. Επαρκεί αυτό για να δείξει ότι υπάρχει το πολιτικό αίτημα, η διεκδίκηση να γίνει αυτό. Και δεν δικαιολογείται απλά, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στους πολίτες, στους ψηφοφόρους, ότι υπάρχει τροχοπέδηση από το Συμβούλιο ενάντια στη βούληση της Ευρωβουλής όταν 12 φορές η Ευρωβουλή έχει ζητήσει να αποτροχοπεδηθούν τα θέματα ε, αυτής της οδηγίας ε, στο, από του Συμβουλίου. Ξέρω σε σχέση με τον Οκτώβριο θα έχουμε και την περίοδο στην οποία θα, θα ξεκινήσουμε σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Ξέρω ότι δεν είναι οι Γερμανοί οι μόνοι οι οποίοι ε, δημιουργούν πρόβλημα σε σχέση με αυτήν την οδηγία Παρόλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι αυτό ίσως καταφέρει να κάνει τη διαφορά και θέλω να πιστεύω ότι όταν θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γερμανίας ίσως αυτό ελπίζω, ίσως να μπορέσει αυτό το θέμα να προαχθεί. Αλλά δεν ξέρω, το ελπίζω. Θέλω να υπενθυμίσω αν δεν γίνει αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε μια εκστρατεία για τις ευρωεκλογές προσπαθώντας να δώσουμε την εντύπωση στους πολίτες μας ότι τους εκπροσωπούν οι ευρωβουλευτές, τους εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δεν μπορεί να επιλύσει αυτό το πρόβλημα, διασφαλίζοντας την ισότητα σε όλα τα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επιθυμούν οι πολίτες. Σε σχέση με αυτό το θέμα θέλω να επαναλάβω τη δέσμευσή μου να καταβάλω κάθε προσπάθεια να εγκριθεί αυτό ώστε το Ευρωκοινοβούλιο να αποτελεί μέρος και τμήμα αυτών των διεργασιών και να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να επιληθούν τα προβλήματα, να επιληθούν τα τεχνικά προβλήματα. Πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση γι' αυτό, μια ανοιχτή διαβούλευση και πρέπει να βρούμε τις σωστές λύσεις για τα θέματα που εκκρεμούν. Δεν αρνούμε ότι εκκρεμούν, αλλά πρέπει να βρεθούν λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό όμως εγκριτό και παραβίστο και κλεισμένο των θυρών με τον τρόπο που ακολούθησε το Συμβούλιο μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. You ask for floor. Ε, thank you, President. And, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ασχοληθεί με τα ζητήματα των ομοφο... ομοφιλοφίλων, των λεσβιών, των αμφιφιλικών και για τα ζητήματα των μειονοτήτων. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ε, μια κατάσταση ντροπιαστική. Θέλω να συγχαρώ την Ιρλανδική Προεδρία για την τεράστια προσπάθεια που έχει καταβάλει ε, για να προωθηθεί αυτός ο φάκελος. Έχουμε συνεργαστεί με τους προσώπους της Ιρλανδικής Προεδρίας στο Δουβλίνο βρισκόμουν την προηγούμενη Παρασκευή και διαπίστωσα την τεράστια πρόοδο που έχει γίνει και πόσο, έχει, ε, πόσο έχουν προχωρήσει τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Ιρλανδία παρά την τεράστια οικονομική κρίση και αυτό είναι εντυπωσιακό και πρέπει να μας διδάξει όλους τι μπορεί να γίνει όταν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση. Νομίζω σωστά τίθεται το θέμα. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Η Γερμανία τα έχει λύσει τα προβλήματα σε τεχνικό επίπεδο και είναι η Γερμανία η οποία μπλοκάρει το θέμα στο Συμβούλιο. Άρα η πικρή πραγματικότητα είναι ότι έχουμε 27 κράτη-μέλη τα οποία ορισμένα από αυτά κρύβονται πίσω από τη Γερμανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή η αλλαγή της κυβέρνησης μας γύρισε προς τα πίσω γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση χωρίς κανένα δισταγμό ε, υποστήριζε ιδιαίτερα τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τώρα με μια κυβέρνηση συνεργασία στην οποία συμμετέχουν και οι φιλελεύθεροι έχουμε ε, πλήρη αλλαγή πορείας. Για να υπάρχει λοιπόν μια δημοκρατική διαδικασία πρέπει όχι μόνο οι ψηφοφορίες αλλά και οι συζητήσεις του Συμβουλίου να είναι δημόσιες έτσι ώστε να μπορούν να λογοδοτούν στα εθνικά κοινοβούλια στους Ευρωπαίους πολίτες, ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα τόσο θεμελιώδες όπως τα δικαιώματα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια οικονομική συνεργασία. Είναι, ένας, ε, είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από όλα αυτά που μάθαμε ε, από την πρόοδο που σημειώσαμε όταν καταλάβαμε ότι θα πρέπει να προασπίζουμε τα, τα, τα δικαιώματα και βρισκόμαστε σε μια, σε μια κατάσταση στην οποία προχωρούμε με τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Συγκρίνεται το με το τι γίνεται για την οικονομία. Έχουμε συνέχεια συνόδους επί συνόδων για τα οικονομικά θέματα, ενώ για τα θεμελιώδη δικαιώματα συγκρίνετε το τι γίνεται, απλώ στέλνουν κάποιου διπλωμάτες σε κρυφές συναντήσεις στις Βρυξέλλες που δεν καταλήγουν σε συμπέρασμα. Οι πολίτες θα κρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από το κατά πόσον τηρεί τι αρχέ τη. Ετέθη το θέμα του κατακαιρμανισμού των οδηγιών. Σας προειδοποιώ και απευθύνομαι και προς την Επιτροπή σας και στο Συμβούλιο σας προειδοποιώ μην τολμήσετε να δημιουργήσετε μια ιεραρχία, μια ιεράρχηση της ε, καταπίεσης τελικά. Ακριβώς αυτό προσπαθούσε να κάνει η Επιτροπή Μπαρόζο πριν να φέρει αυτή την πρωτοβουλία και συνάντησε την πλήρη αντίδραση, αντίσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από όλες τις πολιτικές ομάδες. Γιατί αυτό τι είναι στην πραγματικότητα, είναι ένας τρόπος να δώσουμε περισσότερα δικαιώματα σε αυτούς που ήδη έχουν και οι ήδη καταφρονεμένοι να γίνουν ακόμη περισσότερο. Η οδηγία αυτή αναφέρεται σε πολλά μορφές διακρίσεων. Με βάση τη θρησκεία, με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό, με βάση την αναπηρία. Αυτό είναι θέμα που θα έπρεπε να είναι στην καρδιά των επιδιώξεών μας. Νομίζω βλέπετε το πάθος με το οποίο υπερασπίζομαι αυτό το θέμα. Πρέπει να έχει κάποια σχέση με το γεγονός ότι είμαι από την Ιρλανδία και τα έχω βιώσει αυτά και ταυτόχρονα έχω και Ισπανούς ε, γονείς. Καλός συνδυασμός. Εάν ε, επιλεγεί η λύση του Υγεία, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Με την οικονομική κρίση έχουμε τερα... τραυμακτικές επιπτώσεις στο κοινωνικό επίπεδο. Βλέπετε ότι ψάχνουμε από διοπομπαίους τραγούς δεν έχω δουλειά, δεν μπορώ να έχω ιατρική περίθαλψη, δεν, ε, δεν μπορώ να πληρώσω το, δίκαιο, το, το δάνειό μου για το σπίτι και ψάχνω να βρω κάποιον να κατηγορήσω. Ψάχνω να βρω έναν αποδιοπομπαίο τράγο και ποιον θα βρω, το μετανάστη, αυτό που είναι ανάπηρο, αυτό που έχει οποιοδήποτε, ε, ε, υφίσταται οποιοδήποτε μορφής διάκρισης. Εξετάζουμε το, στο πλαίσιο του παρατηρητηρίου θεμελιωδών δικαιωμάτων την ομοφοβία διαβάστε την έκθεση. Εάν ακόμα χρειάζεστε να διαβάσετε κάτι για να πιστείτε, διαβάστε το σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ρωσικά. Συμπληρώθηκε ένα ερωτηματολόγιο και διαπιστώσαμε ότι ακόμα και σε πρωτεύουσες οι οποίες υποτίθεται ότι είναι φιλικές προς τους ομοφιλόφιλους, το Παρίσι ή το Άμστερνταμ, οι άνθρωποι αυτοί υφίστανται επιθέσεις βίαιες επιθέσεις και αναγκάζονται να κρύψουν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Γιατί η ομοφοβία προελάβνει. Και γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί οι καλές μας κυβερνήσεις δεν κάνουν... Οι καλές κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα και οι κακές κυβερνήσεις, εκείνες που αδιαφορούν για το θέμα, καταφέρνουν να περάσουν τη θέση τους. Η σιωπή είναι συνενοχή σε αυτές τις περιπτώσεις. Ε, εσείς στην Ισπανία κύριε Πρόεδρε έχετε τις εμπειρίες του εμφυλίου πολέμου. Η Ευρώπη τα έζησε αυτά από το 1938 στο 1945. Ευχαριστώ κύριε Κάσπαν. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ όπως και πολλοί συνάδελφοι ε, ε, ε, γοητευθήκαμε από τον το λόγο σας. Ωστόσο μακρηγορήσατε και θα πρέπει να κλείσουμε το θέμα γιατί έχουμε και το ζήτημα της Frontex να συζητήσουμε μετά. Γι' αυτό θα ζητήσω από τους συναδέλφους να τηρούν το χρόνο. Και οι συνάδελφοι είναι οι εξή. Κυρία Ένστ πρώτα απ' όλα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πραγματικά είναι χρεοκοπία για την πιστοποιητικό χρεοκοπία για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πολλά αυτά χρόνια για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπάρχει ακριβώς σε μια φάση όπου λένε οι πολίτες ε, ότι μεγάλες παρεμβάσεις υπέρ της ελευθερίας τους και υπέρ της ζωής τους κατά κάποιο τρόπο υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια σε σχέση με αυτή τη θέση και ενάντια σε σχέση με αυτή τη συζήτηση. Τι απορρέει δηλαδή για μένα. Για ποιο λόγο εγώ ο πολίτης έχω τόσο μικρό όφελος από όλα τούτα. Και ως Ευρωπαία συνειδητά πρέπει να το, δω, να το δω αυτό. Όταν Πέντε χρόνια βλέπω ότι κάνουμε προσπάθεια γύρω-γύρω να προχωρήσουμε και δεν προχωράμε. Ε, αυτό είναι πιστοποιητικό απόλυτη χρεοκοπία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτονόητο είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από τα χέρια μα και θα χρησιμοποιήσουμε και την εκλογική εκστρατεία, όχι εφέτο αλλά και του χρόνου. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταδείξουμε πού ακριβώ βρίσκεται το πρόβλημα. Και, αν, και όταν στη Γερμανία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή από το Ομοσπονδιακό, Ομοσπονδιακό Γερμανικό Δικαστήριο εξετάζονται θέματα και προχωρούν θέματα για την ισότητα μέσα στο πλαίσιο μιας ε, ε, συμβίωσης ε, και του γάμου, τότε είναι αναγκαίο και πιέζει αυτό. Μια και το συνταγματικό δίκαιο, το σύνταγμα στη Γερμανία το δείχνει σαφώς ότι πρέπει να γίνουν βήματα προς τα εμπρός. Να είμαστε όμως αντιπαραγωγικοί και να κάνουμε το αντίθετο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι τότε θετικό για τις ευρωεκλογέ. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να αξιολογήσουμε αυτή την κατάσταση στις ευρωεκλογέ και να δείξουμε ποιο ρόλο διαδραματίζει η Γερμανία μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ επί της ουσίας να πω τίποτα περισσότερο παρά μόνο ότι είναι σκανδαλώδης αυτή η κατάσταση. Όταν ξέρουμε ότι στη Γαλλία μυριάδες κατέβηκαν σε διαδηλώσεις κατά της, ε, ε, του γάμου ομοφιλοφίλων. Όταν ξέρουμε ότι ξυλοκοπούνται στην Πολωνία και αλλού οι ομοφιλόφιλοι όταν ε, ομολογούν ότι είναι ομοφιλόφιλοι. Όλα αυτά τι βλέπουμε. Συμβαίνουν και βλέπουν κάποιοι πώς ε, για παράδειγμα ξυλοκοπούνται και προπυλακίζονται ομοφιλόφιλοι γιατί διεκδικούν κάποια δικαιώματα με τις ε, διαμαρτυρίες και εκδηλώσεις τους. Αν δεν δράσουμε εδώ πρέπει να πω ότι είναι έσχος. Θα είναι ντροπή για μας ε, και πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε. Thank you, thank you for that. Now, let's short... Ευχαριστώ πολύ. Μία σύντομη απάντηση της ε, Ιρλανδικής Προεδρίας μετά από τα παθιασμένα λόγια που ακούστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Παρακαλώ. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά που άκουσα, αλλά εκπροσωπώντας το Συμβούλιο το μόνο που μπορώ να πω είναι να ξαναπώ ότι ε, χρειάζεται, απαιτείται για την οδηγία αυτή ομοφωνία και επομένως δεν, ε, μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε ομοφωνία. Υπάρχουν ακόμα κάποιες ε, τεχνικές ε, λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν ακόμα στο κείμενο και χαίρομαι που συμφωνεί με αυτό και ο εισηγητής. Ε, ενδεχομένως να συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω αλλά ε, πάντως μπορώ να σας πω ότι ε, ε, στη δικιά μας Ιρλανδική Προεδρία εμείς είδαμε μονάχα τεχνικά ζητήματα, κυρίως όσον αφορά την εκπαίδευση και την κοινωνική ασφάλιση. Δεν έγινε καμία ιεράρχηση των παραβιάσεων και της έλλειψης ισότητας ή της διακριτικής μεταχείρισης. Εκπαίδευση και κοινωνική ασφάλιση. Αυτό μας απασχόλησε και ε, σε σχέση με τις αρμοδιότητες που έχουν τα κράτη-μέλη και τις αρμοδιότητες που έχουν κρατηθεί σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτά μας απασχόλησαν. Επίσης, ένα τελευταίο που θέλω να ξαναπώ. Υπήρξαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες με το κείμενο, πρέπει να βελτιωθούν πριν κατά την άποψή μας ε, καταστεί δυνατόν να ε, θέσουμε το κείμενο υπόψη των ε, αρμοδίων υπουργών έτσι ώστε να ληφθεί η πολιτική απόφαση. Αυτή είναι και η άποψη της Κομισιόν. Νομίζω ναι, αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος να επανέρχουμε στον εισηγητή Ρωμένο. Όχι, δεν θέλει να πάρει το λόγο. Τα άκουσα όλα προσεκτικά και θα τα λάβει υπόψη του. Τελευταίο σημείο της ημερησία διατάξεως για σήμερα το πρωί. Frontex. Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση Επιχειρησιακή Συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της, των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δηλαδή ο οργανισμό Frontex. Υπενθυμίζουμε ότι αναθεωρήθηκε το 2011 η εντολή της Frontex ε, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε ώστε να ληφθούν υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα έχουμε Λέμε λοιπόν ότι ο υπεύθυνο των πολιτικών δικαιωμάτων θα πρέπει ε, να συνεπικουρείται από έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων κτλ. Έχουμε εδώ υπεύθυνο, ε, τον υπεύθυνο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την υπεύθυνο μάλιστα, την κύρια την κυρία Αρνάεθ και έχουμε επίση και τον εκπρόσωπο του Συμβουλευτικού Φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε του δύο συμπροέδρους, τον κύριο Στέφαν Κέσσερ και τον κύριο Αδριάνο Σιλβέστρη. Το 2012 ξεκίνησε η θητεία τους. Τους καλέσαμε λοιπόν για να παρουσιάσουν τα πεπραγμένα των μερικών μηνών δραστηριότητας ε, που ε, προσμετρούν. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Αρνάεθ να μας δώσει την δικιά της αξιολόγηση του έργου ε, της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα δώσω το λόγο στον κύριο Κέσσερ. Κυρία Αρνάεθ, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Είναι μεγάλη τιμή να μπορώ να προσφωνήσω τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ΛΥΜΠΕ σήμερα εδώ. Αυτή η πρόσκληση να σας προσφωνήσω δείχνει ότι τα δικαιώματα μεταναστών υπό τη σημερινή κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό μέλημα και ανησυχία σας. Και συμμερίζομαι πολύ αυτό το μέλημα και την ανησυχία σας, διότι στεναρά πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντίφαση μεταξύ ελέγχου στα σύνορα και θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αλλού. Το Συμβουλευτικό Φόρουμ και εγώ ως αξιωματούχος έχουμε θέσει βάρος σε αυτή την ε, τοποθέτηση όσον αφορά την, το να τονίσουμε τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε από κοινού στη συνεδρίασή σας σήμερα και αυτό ελπίζω ότι θα καταδεικνύει σαφώς πώς συμπληρώνουμε ημέν τους δε στην δράση μας. Ως υπεύθυνοι για την υπηρεσία δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως εσείς σωστά αναφέρατε, ήταν η σύντομη αυτή περίοδος παρόλα αυτά μια περίοδος έντονης δράσης και αυτό ε, θέτει την ε, τροχιά και την κατεύθυνση για το μέλλον η συνολική αρμοδιότητα αυτού του αξιωματούχου του αξιώματος μας είναι να διασφαλίσουμε το να λαμβάνονται υπόψη οι πτυχές για το σεβασμό των δικαιώματων των, του ανθρώπου κάνοντας παρατηρήσεις σε σχέση με τα πιλωτικά σχέδια και της Frontex συνεισφέροντας ένα αποτελεσματικό μηχανισμό εποπτείας των δικαιωμάτων του ανθρώπου με τακτές εκθέσεις και δραστηριότητες εποπτείας της Frontex με επισκέψεις ταυτοποιώντα και εντοπίζοντας ε, ανάγκες ή ελλείψεις ε, και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για αντισταθμιστικά διορθωτικά μέτρα για τέτοιου είδους δράσεις. Γενικά λοιπόν συνεισφέρω σε όλα τα θέματα που αφορούν ε, τον οργανισμό μας για ε, τα δικαιώματα του ανθρώπου. Το πλαίσιο μπορεί να επεκτείνεται σε όλες τις δραστηριότητες ε, που πρέπει να είναι συμβατές με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Διεθνές Δίκαιο και με τη Σύμβαση της Γενέβης του 1951 και τις υποχρεώσεις για προστασία σε διεθνές σε παγκόσμιο πλαίσιο. Η Frontex έχει αναλάβει συγκεκριμένα διαβήματα ώστε να διασφαλίζει ότι αυτές οι υποχρεώσεις ε, με αποτελεσματικό τρόπο θα εφαρμόζονται και θα αποτελούν πραγματικότητα. Για την στρατηγική μας ε, για τα δικαιώματα που υιοθετή, εγκρίθηκε το 2011 αποτελεί σημαντικό θεμέλιο για το έργο μου, η δυνατότητα να αξιολογούνται τα θέματα αυτά και οι επιπτώσεις τους όσον αφορά και την κατάρτιση και εκπαίδευση όλων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Frontex και ευαισθητοποίησή τους Δεύτερον, όλο και περισσότερο συμμετέχουν αυτά τα θέματα και εντάσσονται στο λειτουργικό πλαίσιο της Frontex. Ζητήσαμε να διασφαλίζεται ε, κατάρτιση και ε, κατευθύνσεις σωστές που θα διασφαλίζονται όσον αφορά και τα θέματα ασύλου και την προστασία όσον αφορά μετανάστες σε όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να διασφαλίζονται οι βασικές ανάγκες ε, των μεταναστών, προτού οποιασδήποτε δράσεις αναλαμβάνονται, ώστε να μπορούν στις δράσεις αυτές ε, να ε, καλύπτονται αυτά επαρκώς. Και Όλα αυτά αναφέρονται σαφέστατα στα κείμενα των λειτουργικών δράσεων και σχεδίων. Μία από τι κυριότερε προτεραιότητε όσον αφορά το 2013 είναι η υποστήριξη ενό αποτελεσματικού συστήματο εποπτεία όσον αφορά παράπονα και ε, προβλήματα που ε, αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Δεν είμαστε ένα σύστημα ε, εποπτείας, αλλά ένα μέσο, ένα εργαλείο για τη διασφάλιση αποτελεσματικής εποπτείας, προτείνοντας προτάσεις, συγκεκριμένες λύσεις ε, και διαβήματα που πρέπει να αναλαμβάνονται ότι όταν κάτι πρέπει να επιληθεί. Ο μηχανισμός ε, βασίζεται σε ένα σύστημα ε, λογοδότησης και εκθέσεων και η Frontex παράλληλα υιοθέτησε ένα δεοντολογικό κώδικα για όλους όσους συμμετέχουν στις δραστηριότητες ε, υπό το συντονισμό της Frontex, διατάξεις για το σεβασμό και προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και διεθνές, διεθνείς διατάξεις όσον αφορά την προστασία τους ε, με συμμετοχή και υποχρέωση όλων όσων συμμετέχουν για την αναφορά παραβιάσεων ή παραβάσεων. Όταν έχουμε κάποια αναφορά για παραβίαση ή παράβαση υπάρχει εσωτερικά διεργασία ακολουθείτε για την ε, αντιμετώπιση, αξιολόγηση και επανόρθωση αντιστάθμιση και είμαστε, συμμετέχουμε σε σχέση με αυτές τις διαδικασίες και λαμβάνεται απόφαση για την ε, συγκεκριμένη δράση. Έχουμε λοιπόν ε, και την, ε, το θέμα της εποπτείας και ανάλυσης τέτοιων γεγονότων κατά την αξιολόγηση συμβάντων και προτείνονται λύσεις που πρέπει να δοθούν σε περίπτωση παραβιάσεων ή παραβάσεων και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης υπαλλήλων της Frontex που όχι μόνο αφορούν εσωτερικά τους υπαλλήλους και τα στελέχη της Frontex όσον αφορά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και όσον αφορά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς ε, των όσων συμμετέχουν υπάρχει ευαισθητοποίηση και κατάρτιση για τα δικαιώματα του ανθρώπου και πρόσφατα ολοκληρώνουμε ένα εγχειρίδιο για την κατάρτιση για τους συνοριοφύλακες ε, όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου με ένα ευρύτερο τέτοιο πλαίσιο προσεγγίζουμε όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Πώς ε, αντιμετωπίζω τώρα τον ρόλο μου σε σχέση με αυτά διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες ε, που παρατήρησα κατά τη διάρκεια αυτών των, των δράσεων θα καλύπτονται με τον ε, πιο ενδεδειγμένο τρόπο και με την κατάρτιση και με τις δράσεις μας. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις και το έργο που πρέπει να επιτελεστεί, αλλά η Υπάρχει εδώ και υπάρχουν οι κανονιστικές διατάξεις ε, που παράλληλα με τα θέματα μετανάστευσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη. Θέλω να αναφέρω κάποια πολύ ευαίσθητα θέματα όσον αφορά τις δράσεις ε, Frontex, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, δράσεις στην θάλασσα, στα πελάγη που είναι σε ένα δυσχερέστατο πλαίσιο όσον αφορά τους μετανάστες που καταβάλουν προσπάθεια να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον και για τα θέματα που από κοινού προσπαθούμε στις Βρυξέλλες να ολοκληρώσουμε ένα ε, κοινό δεοντολογικό κώδικα που θα διασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο προδιαγραφών ε, από πλευράς ε, διεργασιών που θα ακολουθούνται και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τεράστιες προκλήσεις που μπορούν να συνοψιστούν στην εφαρμογή του συστήματος ε, εποπτείας με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο, διαθέτοντας έγκαιρα πληροφορίες ε, ώστε να μπορούν ε, άμεσα να αναλυθούν αντισταθμιστικά μέτρα. Καλύτερες διεργασίες για την καλύτερη προστασία ατόμων που περνούν τα σύνορα και έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και τους όσους εμπλέκονται σε αυτό το πλαίσιο για τις ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων, των ανηλίκων, των, σε σχέση και με τους ετούντες άσυλο γυναικών παιδιών στην Ελλάδα σε σχέση με την δυνατότητα βελτίωσης του εσωτερικού ε, δυναμικού για την ε, καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, βελτιώνοντας ε, το δυναμικό των ατόμων που διασφαλίζουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές, έχουν την υποστήριξή μου και είμαστε στη διάθεσή τους να τους συνδράμουμε και φυσικά και για τις άλλες υπηρεσίες και οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, συμμετέχουν σε αυτό το πλαίσιο και από πλευράς ε, διεθνών ε, οργανισμών και φορέων για την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου συνεργαζόμαστε και με αυτούς. Προσβλέπω στα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για την βελτίωση των μεταναστών, τις θέσεις των μεταναστών όσον αφορά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιδόσεις της Frontex μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είναι σαφώς υποχρέωσή μας να συνεισφέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θα ξεκινήσουμε τον κύριο Σιλβέστρη του Συμβουλευτικού Φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καθημέρα σας ε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, ΛΥΠΕ, αξιότιμα πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ έτσι ώστε να κάνουμε μια αναφορά σε σχέση με την εργασία του Συμβουλευτικού Φόρουμ. Πριν δώσω το λόγο στον ε, Στέφαν Κέσλα, τον συναδελφό μου, που ασχολείται με θέματα τράφικινγκ, θα ήθελα να κάνω γενική φύσεω παρατηρήσεις όσον αφορά το Συμβουλευτικό Φόρουμ που εκπροσωπούμε εδώ. Από πλευράς ε, υπηρεσίας θεμελιωδών δικαιωμάτων θεωρούμε το Συμβουλευτικό Φόρουμ ένα σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όχι μόνο σε σχέση με την Frontex, αλλά εν γέννη στα εξωτερικά σύνορα το συμβουλευτικό ε, φόρουμ συνεπικουρεί όχι μονάχα την Frontex αλλά και την ε, διαχειριστική επιτροπή της ε, Frontex στην οποία συμμετέχουν και οι συνοριοφύλακες και άλλοι οργανισμοί. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο λοιπόν. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω είναι το εξής. Η κατάσταση ε, στα εξωτερικά σύνορα είναι προτεραιότητα και για την υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων και για το συμβουλευτικό φόρουμ είτε χερσαία είτε θαλάσσια σύνορα. Ε, πρέπει να σας πω ότι μαζί με το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουμε δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο όσον αφορά ε, την, ε, τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο και όσων διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ε, και βεβαίως ε, ε, σαν υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υπηρεσία μάλλον θεμελιωδών δικαιωμάτων η ΦΡΑ στηρίζει την Frontex γενικότερα. Θεωρούμε ότι εδώ έγκυται και το επικοδομητικό στοιχείο της παρουσίας του Συμβουλευτικού Φόρουμ γιατί μπορεί μπορούμε να δώσουμε ε, στο, στην Frontex τις δεξιότητες, τεχνογνωσίες και πραγματογνωμοσύνη μας έτσι ώστε να καθορίσει ένα καλύτερο τρόπο ε, ε λειτουργίας. Και εμείς με τη σειρά μας βεβαίως ε, έχουμε και το input το, της κοινωνίας των πολιτών και της πλατφόρμας του Συμβουλευτικού Φόρουμ. Θεωρούμε ότι η δημιουργία του Συμβουλευτικού Φόρουμ είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα δώσω τώρα το λόγο στον Στέφαν για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά ε, με τα όσα έχουν ήδη γίνει και τα όσα θέλουμε να πράξουμε στο μέλλον. κύριος Κέσλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που καλέσατε τους συμπροέδρους ε, του Συμβουλευτικού Φόρουμ ε, στην συνεδρίαση αυτή. Ε, θεωρούμε, την εκλαμβάνουμε μάλλον, <clears throat> την πρόσκληση αυτή από πλευρά της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ σαν ένα σημάδι αναγνώρισης της σημασίας που έχει το Συμβουλευτικό Φόρουμ στην προσπάθεια επίλυσης των συστημικών προβλημάτων. Δεν θέλω να μπω τώρα σε διαδικαστικές λεπτομέρειες και να σας κουράσω. Θα ήθελα όμως να ασχοληθώ με ορισμένα θέματα τα οποία μου φαίνονται σημαντικά. Το 2011 τροποποιήθηκε η, ε, ο κανονισμός της Frontex και παρευλήθη ένα νέο άρθρο το οποίο αποτελεί και τη νομική βάση ε, για την ίδρυση του συμβουλευτικού μας ε, φορέα. Ε, αυτή τη στιγμή ε, ε, έχουμε και δύο άλλες ε, υπηρεσίες, την ΦΡΑ και την, το, Συμβουλευτικό Φορέα, που συνεπικούν την Frontex. Το 2013 εστιαστήκαμε σε τέσσερα κεντρικά σημεία. Πρώτον, κάναμε σύσταση για την δημιουργία ενός προσχεδίου κώδικα συμπεριφοράς και καλών πρακτικών. Επίσης, περαιτέρω ανάπτυξη των συστάσεων του ε, μηχανισμού. Τρίτον, ε, εκπαιδευτικό υλικό, υλικό κατάρτισης. Τέταρτον, έρευνα σχετικά με την ε, πληροφόρηση ε, σε σχέση, με καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, τρόπους επίλυσης διαφορών. Πρέπει να σας πω πάντως ότι συνειδητοποιούμε ότι ούτε εμείς ούτε και η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορεί να λύσει τα διαρθρωτικά προβλήματα το φόρουμ δεν μπορεί, δεν είναι σώμα που λαμβάνει αποφάσεις, μπορεί όμως να κάνει συστάσεις. Δεν μπορεί από μόνο του ε, να ξεκαθαρίσει ε, ασάφιες Ε, αλλά μπορεί να κάνει κάποιες προτάσεις ε, είτε στην Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είτε στις εθνικές, ε, στα, εθνικά σώματα τα οποία ασχολούνται με το θέμα αυτό. Δηλαδή που ασχολούνται με τη φύλαξη των συνόρων. τα, έχουμε τον, ε, ε, ε, την ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών που ανέφερε και παραθέτω ε, η διαχείριση των ε, ε, συνόρων της Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ακόμα επιτύχει το βέλτιστο βαθμό αλλά γίνονται καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες. Το Συμβούλιο της Ευρώπης επίσης αναφέρεται σε πολύ, κάποιες πολύ συγκεκριμένες συστάσεις μία εκ των οποίων είναι ε, να ενισχυθεί η δημοκρατική λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι και ο υπεύθυνο μελιδών δικαιωμάτων και το Συμβουλευτικό Φόρουμ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ε, να αναφέρονται απευθεία στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το λάβετε υπόψη σα. Επίση, ε, μπορούμε να κάνουμε συστάσεις στην Frontex σχετικά με το τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήδη ο Συμπρόεδρος ανέφερε ότι και η Υπηρεσία Θεμελιδών Δικαιωμάτων ε, ε, κάνει συστάσεις ε, όσον αφορά την προστασία των συνόρων στη Μεσόγειο. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι ο ρόλος της Frontex έχει ξεπεράσει τον απλό συντονιστικό ας πούμε ρόλο, τον, τον συντονισμό δηλαδή μεταξύ των δραστηριοτήτων των κρατών μελών αλλά λαμβάνει υπόψη και τον ε, ενωσιακό και το διεθνή νόμο για τα νομοθεσία διεθνή και ενωσιακή για τα ανθρώπινα ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Ο κανονισμός της Frontex δίνει στην υπηρεσία ε, την δυνατότητα κοινών επιχειρήσεων και ε, υποχρεώνει την καταγραφή συστημικών ε, ε, παραβιάσεων καθώς επίσης και την, δίνει τη δυνατότητα άρνησης της χρηματοδότησης κάποιων δραστηριοτήτων ή επιχειρήσεων σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς όμως να παρέχει και ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο για την κατάσταση αυτή. είναι κοινά συμφωνημένο ότι ε, θα πρέπει όλες ε, οι δραστηριότητες της Frontex ε, να διασφαλίσουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός διασφάλισης της εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας ούτε υπάρχουν πρόνοιες οι οποίες να προβλέπουν κοινό μηχανισμό προσφυγής έναντι ε, κρατών που συμμετέχουν σε κοινέ ε, δράσεις ε, και επιχειρήσεις. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Από τη στιγμή που οι καταγγελίες δεν μπορούν να προχωρήσουν κανονικά βάσει αρμοδίων οργάνων το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο και κυρίως η δική σας ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσει ενδελεχώς την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημιουργήσει αυτούς τους, στρατηγικού αυτούς τους στρατηγικούς όρους και προϋποθέσεις που αποτελεσματικά θα προστατέψουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ε, θα πρέπει να ελέγχεται από το κατά πόσον εφαρμόζει τις αρχές που η ίδια έχει εξαγγείλει. και επίσης θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω συμφωνίες ανάμεσα στην Frontex και ε, τρίτες χώρες. Η κατάσταση στο Μαρόκο ας πούμε ε, είναι καταστροφική. Παρ' όλα αυτά ε, οι Ισπανικές αρχές και οι Ισπανοί συνοριοφύλακες στενά συνεργάζονται με την Frontex όσον αφορά την επανεισδοχή. Συγγνώμη που δίνω σαν παράδειγμα ενώπιόν σας το παράδειγμα των Ισπανών συνοριοφυλάκων. Εν πάση περιπτώσει περιπτώσει όμως. Εμείς πρέπει να ζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή Λίμπε να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ του εκπροσώπους του Συμβουλευτικού Φόρουμ και την εκπρόσωπο, την αρμόδια για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τώρα θα ήθελα να γνωρίζω αν κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να λάβουν το λόγο. ξεκινήσουμε από τον κύριο Ο κατάλογος των ομιλητών έχει τουλάχιστον 6 ομιλητές και πρέπει να σας ενημερώσω ότι έχουμε 30 λεπτά στη διάθεσή μας. Άρα προσπαθείτε να μην γρηγορείτε. Κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ και θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για το έργο τους και για τις παρουσιάσεις τους. Νομίζω ότι έχουμε μια μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσουμε εδώ και είναι κάτι που το συζητάμε συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απ' τη μια επιθυμούμε τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των επικών τρίτων χωρών που έρχονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των σύνορων. Εάν κανείς διαβάσει τις εκθέσεις αξιολόγησης του συστήματος Σέγγεν, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν κενά στην ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, άρα η πρόκληση είναι μεγάλη. Όταν επιδιώκουμε να ε, εξισορροπήσουμε αυτές τις δύο επιδιώξεις και να ε, ανταποκρινόμαστε και στις δύο Πρώτο μου ερώτημα λοιπόν έχει σχέση με την κατάρτιση των συνοριοφυλάκων. Είπατε ότι δεν έχετε την αρμοδιότητα να συμμετέχετε τάσχεται στις καταρτήσεις των συνοριοφυλάκων. Βεβαίως οι συνοριοφύλακες οι οποίοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις της Frontex αλλάζουν συνεχώς. Άρα χρειάζεται κατά την άποψή μου μια διαρκής προσπάθεια για να είναι αποτελεσματική αυτή η κατάρτιση και πρέπει να το δούμε στενά αυτό το ζήτημα. Στο νομοθετικό επίπεδο πάντως, σε όλα τα σχετικά κείμενα, ήμουνα εισηγητής για τις αλλαγές στο δεύτερο πακέτο για τον ε, κώδικα συνόρων. Συμπεριλάβαμε την υποχρέωση κατάρτισης των συνοριοφυλάκων και, και σε άλλα νομικά κείμενα ε, έχουμε εισάγει τέτοιες πρόνοιες. Άρα δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος κάποιο μέλος του Κοινοβουλίου που θα έλεγε ότι δεν είναι ζήτημα προτεραιότητας για εμάς. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την, αυτή την κατάρτιση, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματά σας και πιθανόν να έχετε και πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Δεύτερο ερώτημα. Αναρωτιέμαι αν έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε σε σχέση με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την πλευρά των τρίτων χωρών, γιατί γνωρίζω ότι έχουμε συχνά συμφωνίες επανεισδοχής με αυτές τις χώρες, προσπαθώντας να έχουμε καλύτερη επιχειρησιακή συνεργασία και στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως και σε άλλους τομείς και αναρωτιέμαι εάν ασχολείστε και με αυτή το τομέα, με αυτό το θέμα και αν θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Πώς είναι η κατάσταση ε, για τους ε, παράτυπους μετανάστες οι οποίοι φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα, τι γίνεται με τους διακινητές, τι γίνεται με όλες αυτές τις καταστάσεις που νομίζω όλοι γνωρίζουμε και πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην προσπάθειά μας να σταματήσουμε αυτό πριν να φτάσει στα εξωτερικά σύνορα. Και τέλος, αναρωτιέμαι πώς εξελίχθηκε η κατάσταση, πού βρισκόμαστε δύο-τρία χρόνια μετά από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να ε, εισάγουμε το ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο τομέα αυτό. Έχουμε τη δική σας ε, θέση, τις δικές σας εκθέσεις, ε, τις εκθέσεις της, της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της υπηρεσίας, των Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών για να ρωτιέμαι τελικά υπάρχει βελτίωση, βελτιώνονται τα πράγματα ή όχι. Κατά την άποψή μου, σε νομοθετικό επίπεδο η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Υπάρχετε εσείς έχει δημιουργηθεί το φόρουμ. Ένα φόρουμ που έχει όλες τις ε, δυνατότητες για να προωθήσει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Επίσης έχουν αυξηθεί σημαντικά οι μεταναστευτικές ροές, άρα τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Άρα, με λίγα λόγια, έχει βελτιωθεί η κατάσταση ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επόμενος ομιλητής. Κύριε Σαντιού. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την κυρία Αρνάεφ και τους εκπροσώπους του Φόρουμ για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει για την προστασία των δικαιωμάτων των Ρωμά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Frontex. Το Συμβουλευτικό Φόρουμ και το Γραφείο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν προκειμένου να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των Ρωμά και των μειονοτήτων. Άρα είναι επιφανέ ότι το έργο σας είναι πολύ σημαντικό. Και σας διαβεβαιώνω ότι έχετε την πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή μας πάντα επιδιώκει να προωθεί το σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών. Οι αρμοδιότητες της Frontex έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά όταν αυξάνονται οι αρμοδιότητες αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Για παράδειγμα η Frontex βρίσκεται στο κέντρο του νέου συστήματος διαχείρισης του συνόρων, το Eurosur, που προωθείται. Και δώσαμε σε αυτό το νέο σύστημα και αυξημένες αρμοδιότητες σε σχέση με, τις, ε, ε, με τη διάσωση στη θάλασσα. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Δεν γνωρίζουμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη επιτόπου. Και αυτό ε, ε, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εσάς, από την πίεση που θα ασκηθεί στη Frontex και στους ε, υπαλλήλους της και στους συνοριοφύλακες να σέβονται τα δικαιώματα των μεταναστών, το δικαίωμα στη ζωή, για παράδειγμα. Πιστώνω με χαρά ότι δημιουργήθηκε ο μηχανισμός αξιολόγησης του συστήματος Schengen, και σύντομα θα μας δώσει τα αποτελέσματά του και επίσης είναι ε, ε, θετικό το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται και ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτή την αξιολόγηση, την αξιολόγηση του συστήματος Σέγγεν δηλαδή. Πρόσφατα επίσης υιοθετήθηκε ένα πακέτο νομοθετικό με στόχο την βελτίωση της μεταχείρισης των μεταναστών. Άρα η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο βελτιώνεται η νομοθεσία που προσπίζει τα δικαιώματα των μεταναστών. Αλλά με αυτό κατά νου γνωρίζουμε όλοι ότι άλλο πράγμα είναι νομοθεσία και άλλο πράγμα η πράξη. άλλο πράγμα η πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να αυξηθεί, να μεγαλώσει αυτό το χάσμα. Θέλουμε στην πράξη τα δικαιώματα των μεταναστών να διασφαλίζονται, όχι μόνο στα χαρτιά. Και σας ευχαριστώ για το έργο που κάνετε για να γίνει αυτό πραγματικότητα κυρία Μπιγιάμ. Και πάλι υπενθυμίζω να μην, να μην ε, να τηρείτε το χρόνο. Η κυρία Βίξτρο μάλλον πρώτα. Εσείς κύριε Πρόεδρε θα αποφασίσετε, αλλά αν μου δίνετε το λόγο δεν θα πω όχι. Ε, απολογείται ο Πρόεδρος. Εντάξει, αφού η κυρία Λιάμ είναι από την ίδια ομάδα με εσά, δεν έχει σημασία σε ποιον από, τους, τις δυο θα δώσω πρώτα τον λόγο. Υπάρχει μια ιεραρχία στα πάντα, λέει η κυρία Βίξτρομ, έτσι δεν είναι. Τέλο πάντων, έχετε το λόγο. Κυρία Βίξτρομ, σα ευχαριστώ για αυτέ τι αναλυτικέ παρουσιάσει. Τις παρακολούθησα προσεκτικά. σκιώδη, ήμουν σκιώδης στη για τη νέα εντολή της Frontex και θεωρώ σημαντικό να παρακολουθεί κανεί ένα ζήτημα όταν ξεκινά να ασχολείται με αυτό. Και ορίζω λοιπόν την παρουσία σα. Θεωρώ ότι ε, συνάδελφοι θα πρέπει να είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να δημιουργηθεί αυτό το συμβουλευτικό φόρουμ, γιατί θυμάμαι ότι, ότι συνεργαστήκαμε καλά με ορισμένους συναδέλφους που δυστυχώς τώρα έφυγαν και καταφέραμε τελικά να δημιουργηθεί αυτό το φόρουμ. μας ε, παρουσίασε το πρόγραμμα εργασιών του για το 2013 το Φόρουμ και το καλωσορίζω, η συνεργασία λειτουργεί. Η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει συνεισφέρει στο πρόγραμμα εργασιών αυτό. Επίσης καλωσορίζω την αποστολή επιτόπου ε, ε, ανθρώπων οι οποίοι θα επιτηρούν την κατάσταση. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και στις περιπτώσεις ε, ε, από, κοινού επιχειρήσεων για επαναπροωθήσεις. Γνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της Frontex και θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον αυτό έχει επηρεάσει το έργο σας και ποιες ήταν οι συνέπειες που πιθανώς να ε, βλέπετε να έχει, έχουν οι αλλαγές στους στη χρηματοδότηση, αν αυτό θα επηρεάσει την ποιότητα. Είναι προφανές ότι όλοι πρέπει να σέβονται όλα τις, όλη την νομοθεσία, τον, τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, σε πρακτικό επίπεδο πρέπει να δούμε πώς γίνονται σεβαστά αυτά. Και θα ήθελα να γνωρίσω ποιες είναι οι συγκεκριμένες συστάσεις σας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν διαδικασίες αποτελεσματικού ελέγχου. Αναρωτιέμαι επίσης εάν υπάρχει δημιουργηθεί ένα σύστημα υποβολής ε, καταγγελιών και πώς αυτές αξιολογούνται. Μια και έχουμε ε, ξεκινήσει τις συζητήσει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ο συγητή είναι ο κ. Κοέλιο, για την νέο κανονισμό για την επιτήρηση των θαλασσίων εξωτερικών συνόρων. Θα ήθελα επίση να γνωρίζω τι προβλέπετε ότι πιστεύετε ότι, ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του Συμβουλευτικού Φόρουμ για αυτόν τον τομέα, σε αυτόν τον κανονισμό. Και τι θα θέλατε να προσπαθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εισάγει στον κανονισμό αυτόν. Ευχαριστώ κυρία Κέλλαρ. Κυρία Κέλλαρ, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και μας κάνατε αυτές τις παρουσιάσεις. Πράγματι εργαστήκαμε σκληρά σε αυτή την κοινοβουλευτική επιτροπή, ώστε τα όργανα σας, οι φορείς σας να μπορέσουν ε, να προαχθούν και να εγκριθούν ε, ε, και το καθεστώς τους και σε σχέση και με τη Frontex και έχουμε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή ιδιαίτερη δέσμευση ώστε η δική σας δουλειά να μπορεί να διευκολύνεται και να είναι δυνατόν να αναπτύσσεται. Επίσης, συμφωνώ ότι δεν θα έπρεπε να υπερβαρύνουμε το έργο σας Προφανώς ε, δεν ε, είσαστε εσείς ε, υπεύθυνοι για τα θέματα των ε, θεμάτων εσωτερικών διακρίσεων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά τα φαινόμενα. Αυτό που μπορείτε όμως να κάνετε είναι να υποπτεύετε και να δίνετε επισημάνσεις και κατευθυντήριες γραμμές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό περιεχόμενο σε αυτό το έργο. Πολύ σημαντικό θέμα. Τρεις ερωτήσεις θα είχα. Πρώτα, συστάσεις. Μπορείτε να υποβάλλετε συστάσεις. υποβάλατε ήδη κάποιες συστάσεις. Αν ναι, ποιες. Και ποια ήταν η συνέχεια των, τις οποίες έτυχαν αυτές οι συστάσεις σας. Δεύτερον, έχετε και αντιμετωπίζετε το θέμα των διαφόρων επιμερισμένων αρμοδιοτήτων, αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών όσον αφορά τις δικές σας δράσεις και τα κράτη-μέλη. Πώς θα έπρεπε αυτά τα θέματα να αντιμετωπίζονται σε σχέση με τα κράτη-μέλη, τους εθνικούς, για παράδειγμα, σύνοριοφύλακες. Το εντάσσετε και αυτό μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και τρίτον, όσον αφορά την συνέχεια και συνεκτικότητα των δράσεων, όσον αφορά για θέματα ε, αδικαιωμάτων του ανθρώπου, την τελευταία φορά που είχαμε συζητήσει για αυτά τα θέματα με τον αρμόδιο που είχε προσέλθει στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή, μας είπε ότι εκπονούσαν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές ή κριτήρια πότε θα εφαρμοζόντουσαν όλα αυτά, πότε θα θεωρεί το κάτι σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ και αρκετό διάστημα υπάρχει λοιπόν αυτό. Και τώρα δεν υπάρχουν τέτοια κριτήρια ακόμα. Δεν έχουν εκπονηθεί. Πώ έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, σε ποια φάση βρίσκονται, τι μπορούμε να κάνουμε για να σα υποστηρίξουμε να προαχθούν περισσότερο. Σα ευχαριστούμε. Ernst, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Η Frontex ανήκει στις, ε, στους προσωπικότατους εφιάλτες μας και επανειλημμένα όταν βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα και δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το όργανο αυτό αλλά κυρίως και με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω ε, για τις εισηγήσεις ε, που μας έγιναν ε, την κυρία, από την κυρία Αρνάτ και τον κύριο Κέσλερ ιδιαίτερα για το σε ποια σημεία βρισκόμαστε και κινούμαστε. Θέλω να πω ειλικρινά γι' αυτό ότι πάντα είναι καλό να έχουμε συστήματα επόπτευσης και εποπτείας. Πάντα είναι καλό να υπάρχουν συμβουλευτικά και διαβουλευτικά όργανα, σίγουρα, εντάξει, αλλά όταν έχουμε τέτοια όργανα πρέπει οι αρμοδιότητες να είναι δεδομένες και διασφαλισμένες. Ο χαρακτήρας συστάσεων που υποβάλλει ένα τέτοιο φόρουμ είναι πενιχρός, είναι πολύ ισχνός για να μπορεί να ικανοποιηθούμε. Ε, τις εξής ερωτήσεις θα είχα να σας διατυπώσω και θα ήθελα συγκεκριμένες χειροπιαστές απαντήσεις προς την κυρία Αρνάευ πρώτα. Τα συστήματα επόπτευσης και εποπτείας. Μιλήσατε για αυτά πιο πριν. Θα ήθελα να μου πείτε ποια αποτελέσματα υπάρχουν. Τι έγινε. Τι ξεκίνησε και ποια είναι η εποπτεία και τα ε, εποπτικά, συστήματα, ποια αποτελέσματα έδωσαν χειροπιαστά. Μπορείτε να μας πείτε κάτι σχετικά. Επίσης είπατε ότι διοντολογικός κώδικας και σεβασμός δικαιωμάτων του ανθρώπου και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σημαντικό είναι να σας αναφέρονται παραβάσεις και παραβιάσεις. Πόσες τέτοιες παραβιάσεις και παραβάσεις σας αναφέρθηκαν και γνωστοποιήθηκαν όσον αφορά την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του ανθρώπου. Προς τον κύριο Κέσλα, κυρίως την εξή ερώτηση θα είχα. Αναφέρεται στην έκθεση, στην έκθεση που συντάξατε. Πόσες δράσεις ε, σε σχέση με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν ποιε συνέπειε. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα που μπορείτε να μα αναφέρετε. Τι συνέβη και τι ήταν σημαντικό για, την, για το πάγωμα, την ανάκληση ή την ε, ε, κατάργηση κάποιων δράσεων. Μα είπατε ότι είναι δυνατόν να υποβάλλονται τέτοια παράπονα. Ποια παράπονα υποβάλλονται, ποια σα υποβλήθηκαν, τι είδου είναι αυτά τα παράπονα. Μπορείτε κατηγοριοποιημένα σε κατηγορίε ε, να μα παρουσιάσετε αυτό το φαινόμενο, αυτό το γεγονό. Κατά τα άλλα η κατάσταση όπω έχει σήμερα με ανησυχεί ιδιαίτερα σε σχέση με το ότι χάνουν τη ζωή του πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλοί μετανάστε όταν προσπαθούν να προσέλθουν στην Ευρώπη, με θλίβει ιδιαίτερα και με συγκλονίζει. Και θα ήθελα αυτή η πτυχή από πλευρά τη Επιτροπή Λίμπε να τύχει συνέχεια εκ του σύνεγγυ. Ευχαριστώ. Now, Madame Guillaume, vous avez la parole. Κυρία Γκυγιόμ, παρακαλώ τώρα, έχει τον λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε. Λυπούμε αν είχατε δώσει κάποια έγγραφα που δεν είχατε δυνατότητα να τα μελετήσω, θα το κάνω μετά. Όπως έλεγε και η Σεσίλια προηγουμένως, ε, ήμουν και εγώ από τις χειώδεις ε, που παρακολούθησαν τα ζητήματα αυτά. Δεν είμαι και δεν έχω την ίδια ιδηλιακή έτσι άποψη για τις διεργασίες, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ ικανοποιητικό που βλέπουμε ότι πλέον υπάρχουν τέτοιου είδους όργανα. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε τώρα στην κατάσταση των συνόρων, να εντείνουμε ε, μια, τον διάλογο με την Frontex που θα πρέπει να ενισχυθεί, αλλά και να δούμε από κοντά τις δικές σας δραστηριότητες είχα τρεις άξονες ε, ερωτήσεων. Πρώτον, θέματα συνεργασίας. Επιμείνετε σε αυτό. Είπατε ότι ε, πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε την ε, συνεργασία. Δεύτερον, πρόσβαση σε δόκιμες πληροφορίες. Πιστεύετε ότι πλέον έχετε τη δυνατότητα να λάβετε αυτές τις πληροφορίες ή πρέπει να ανοίξουν και άλλα πεδία. Τρίτον, κατά την άποψή σας υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, μια ιδιαίτερη ανησυχία που έχετε πάνω στην οποία θέλετε εσείς να εμβαθύνετε τη σκέψη σας και στην οποία εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε ε, και το θέμα των προσφυγών, καταγγελιών, αυτό μας απασχολεί πολύ. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα ακούσαμε και τις απόψεις ε, των ε, ε, βουλευτών. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Προτείνω εν συντομία να απαντήσετε από... Να ακούσουμε λοιπόν και την υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και τους συμπροέδρους. Απλώς να έχετε το νου σας, να μην ξεπεράσετε το χρόνο. Κυρία Αρνάεφ θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο γρήγορα όσον αφορά το θέμα της ε, κατάρτισης. Υπάρχουν αρκετές ε, ε, ικανότητες κατάρτισης και προγράμματα τα οποία λειτουργούν ας πούμε παροχή υλικού που πρέπει να υλοποιήσουν, να εφαρμόσουν άλλοι. Και ήδη από την πρώτη στιγμή ασχολήθηκα με αυτό το θέμα, κυρίως με την κατάρτιση των συνοριοφυλάκων. Όμως ε, τα European Border Guard Teams ε, είναι αυτά τα οποία ασχολούνται και κάνουν την ε, κατάρτιση, αλλά η συνεργασία είναι πολύ καλή. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τα αποτελέσματα. Συνεργασία με τρίτες χώρες. Η Frontex λειτουργεί ε, στο πλαίσιο των, ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Υπάρχουν όμως και διμερείς ε, συμφωνίες οι οποίες αφορούν τεχνικά στοιχεία κυρίως της συνεργασίας και αναφέρονται και σε στοιχεία ανάλυσης κινδύνου, κατάρτιση κτλ για την ώρα δεν έχω δει όλες αυτές τις συμφωνίες και δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Δηλαδή ε, η αρχική μας μέρημνα ήταν να δούμε εντός των συνόρων τι γίνεται και όχι εκτός. Θα το κοιτάξω όμως το θέμα αυτό της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Στο εγγύς μέλλον μάλιστα. Η κατάσταση είναι καλύτερη ή χειρότερη. Με ρωτήσατε. Δεν ήμουν εδώ πριν από τρία χρόνια, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει πρόοδος. Έχω δει προόδους, έχω δει εξελίξεις, έχω δει να εφαρμόζονται καλύτερα συστήματα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει χώρος βεβαίως για βελτίωση. Θα πρέπει να δούμε και πώς θα λειτουργήσει καλύτερα η δική μας συνεργασία να δούμε, δηλαδή να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η συνεργασία, γιατί ένα εξάμεινο δεν είναι αρκετό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για όλα τα λόγια στήριξης που ακούσαμε, τα εκτιμούμε δεόντως. Όσον αφορά τις κοινέ επιχειρήσεις επαναπατρισμού, δεν έχουμε δεν έχω καμία ε, κανένα πρόβλημα και καμία, ε, κανένα περιορισμό στην ε, πρόσβαση των στοιχείων που ζητώ όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Σχετικά με τις συστάσεις, το ανέφερα ίσως πολύ γρήγορα προηγουμένως. Εγώ προσπαθώ να αναθεωρήσω κάποια σχέδια και να κάνω, ε, προς, ε, να κάνω κάποιες προσθήκες ή κάποιες ε, συστάσεις έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά την ολοκλήρωση ή την αναβολή κάποιων επιχειρήσεων, ε, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει συνολικό πακέτο και αυτές τις αποφάσεις τις παίρνει το senior management. τα στοιχεία αυτά αναφέρονται ξεχωριστά. Το σύστημα είναι αυτό που είναι και τα κριτήρια βασίζονται στο, ε, στα φαινόμενα τα οποία είναι σοβαρά ε, ή ε, ε, που επιμένουν ας πούμε ότι είναι καταστάσεις οι οποίες ε, επανέρχονται διαρκώς. Βεβαίως υπάρχει χώρος για βελτίωση των κριτηρίων. Τα ευρήματα, κοιτάξτε, πολύ σχέση έχει και με την ε, διαφορετικότητα των ε, διαφορετικών εντολών, ε, των εμπλεκομένων στις επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο δύσκολο να έχει κανείς πρόσβαση στην πληροφόρηση, αλλά το ζήτημα είναι να διαφοροποιεί κανείς κάποιες υπόνοιες σε σχέση με κάποιες σωστές πληροφορίες οι οποίες μπορούν να καταλήξουν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. για την ώρα μέχρι τώρα έχω λάβει έξι ε, καταγγελίες βάσει υπονοιών ε, για ε, παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχει ξεκινήσει η ανάλυση. Και το ελάχιστο που μπορώ να πω είναι ότι τουλάχιστον ευαισθητοποίηση υπάρχει ε, σε σχέση με καταστάσεις ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, των μεταναστών. Δηλαδή έχει γίνει κατανοητό ότι υπάρχει ένα ζήτημα και νομίζω ότι η κοινή γνώμη και οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι ευαισθητοποιημένοι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αρνάεθ. Κυρία Κέσλερ, εσείς θα μιλήσετε πρώτος. Κοιτάξτε, για να απαντούσα σε όλες τις ερωτήσεις θα έπρεπε να είχα τουλάχιστον μια ώρα μπροστά μου. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Όχι, εμεί δεν έχουμε καμία ανάμειξη στη συνεργασία τη Frontex με τρίτε χώρε. Ούτε στη σύνταξη δημιουργών συμφωνιών. Νομίζω ότι η κατάσταση, ρωτάτε αν η κατάσταση έχει αλλάξει τα τελευταία 14 χρόνια. Κοιτάξτε, έχει βελτιωθεί πολύ το νομοθετικό πλαίσιο. Έχει βελτιωθεί και ο αντίκτυπος αυτής της νομοθεσίας. Παρ' όλα αυτά κρατάω κάποιες επιφυλάξεις. Γιατί έχουμε πολλά ατυχήματα, έχουμε πολλά συμβάντα με νεκρούς, κυρίως στα θαλάσσια σύνορα. Μη λησμονείτε πάντως ότι εμεί ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε το 2013. Ο μιλητή μιλάει εντελώ εκτό μικροφώνου, οι διερμηνεί δυσκολεύονται πολύ να τον ακούσουν. Όλοι προσπαθούν να κάνουν ε, τη δουλειά που ε, έχουν ε, αναλάβει, αλλά μην λησμονείτε ότι πολλά πράγματα πρέπει να τα κάνουμε εκτός ε, της, ε, του, του πλαισίου εργασίας μας ας πούμε και των υποχρεώσεων εργασίας μας. Όπως είπα και θα ξαναπώ και θα λέω διαρκώς, δεν, ε, αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος από το Κοινοβούλιο. Είναι μια πολύ, ένα πολύ σημαντικό εχέγγυο αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις κοινέ επιχειρήσεις της Frontex. ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει ε, αυτή, αυτό το σωστό monitoring, η σωστή εποπτεία που η οδηγία για την επιστροφή και η πανεσδοχή ε, προβλέπει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. επίσης σχετικά με μία ερώτηση. Ξαναλέω, δουλεύ, αρχίσουμε να δουλεύουμε ε, την αρχή του 2013, δεν έχουμε κάνει ακόμα συστάσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ε, συζήτησης ε, με το Senior Management Board, με τα κράτη-μέλη, με την υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν έχουμε κάνει ακόμα συγκεκριμένες συστάσεις. η ερώτηση για τα κριτήρια απαντήθηκε ήδη. Είμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη, κυρίως με το Management Board. Εγώ έχω πάει ε, στις συνεδριάσεις του Management Board, εγώ έχω κάνει κάποιες προτάσεις ε, και άλλες ε, τις υποδέχτηκαν με σκεπτικισμό, άλλες με πιο θετικό τρόπο. δεν έχουμε ακόμα, δεν έχει υπάρξει άρση ε, ε, επιχειρήσεων για την ώρα. Επίσης δεν λαμβάνουμε μεμονωμένες καταγγελίες. Δεν είναι δικιά μας ε, δουλειά για την ώρα τουλάχιστον, επομένως δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση για μεμονωμένες καταγγελίες. Επίσης να σας πω δεν έχουμε την ίδια καλή θέση ως, όπως η υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων να συζητούμε ε, απευθείας με την ε, Frontex και όσον αφορά και την πρόσβαση σε κάποια έγγραφα υπάρχουν, υπάρχουν ακόμα κάποιες εφές ζώνες όσον αφορά την προσβασιμότητα που έχουμε σε έγγραφα. Πρέπει να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Ε, θέλετε να, να μιλήσετε και εσείς κύριε Σιλβέστρη. Ναι, όσον αφορά τις συστάσεις, θα σας δώσω ένα παράδειγμα σχετικά με το ποιο είναι το feedback το οποίο μπορεί να δώσει στην ε, feedback το Συμβουλευτικό Φόρουμ όσον αφορά τον κώδικα συμπεριφοράς ε, για τις ε, επιχειρήσεις επανεισδοχής. Κάναμε καμιά τριανταριά σχόλια. Από τα τριανταριά σχόλια είδαμε ότι τα μισά τουλάχιστον από αυτά ενσωματώθηκαν ε, στις ε, ε, προτάσεις της Frontex. Επομένως υπάρχει, υπάρχει κάποιος αντίκτυπος, αλλά όχι πλήρης. Σχετικά με το εάν έχει υπάρξει βελτίωση ή όχι από τη στιγμή που άρχισε να παρακολουθεί τη εργασία της Frontex από τις υπηρεσίες θεμελιδών δικαιωμάτων και συμβουλευτικό φόρουμ κτλ. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μας έχουν υπάρξει πολλές σημαντικές ουσιαστικές αλλαγές στα χαρτιά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να επικεντρωθούμε έτσι ώστε και στην πράξη και εκεί έξω δηλαδή που λαμβάνει η χώρα η δράση στα εξωτερικά σύνορα να βελτιωθούν τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που με προθυμία δεχτήκατε την πρόσκλησή σα. Ευχαριστούμε γιατί συμμετείχατε σε αυτήν την πολύ καρποφόρα και επικοδομητική συζήτηση. Θα είμαστε εδώ, θα σα παρακολουθούμε, θα βλέπουμε τη δουλειά σα. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 3 το απόγευμα 8 Ιουλίου. Γεια σας.